κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού. Η πρώτη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αφορά την κατάσταση των ε, ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγγάντα. Πριν την έναρξη της συζήτησης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για να ζητήσετε το λόγο με τη διαδικασία Catch the Eye ή για να θέσετε ερώτηση με γαλάζια κάρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον συνηθή τρόπο εγγραφής και το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ να έχετε πάντα μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας. Αν θέλετε να εγγραφείτε για τη διαδικασία Catch the Eye σας παρακαλώ μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα χωρίς να περιμένετε το τέλος της συζήτησης. Το λόγο έχει η κυρία Τσόουνς εκ των συντακτών της ερώτησης. Για ένα λεπτό. Thank Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει διακομματική στήριξη της συζήτηση και του ψηφίσματος ε, Κάτι το οποίο δείχνει ότι αλλάζουν οι νοοτροπίες και οι στάσεις. Είμαστε αλληλέγγυοι σήμερα απέναντι στους γενναίους ε, συνανθρώπους μας, μέλη σεξουαλικών μενοτήτων στην Ουγκάντα, οι οποίοι ε, καταστέλλονται, ε, καταστέλλεται η ίδια η φύση τους από το κράτος. Ζουν υπό τις πλέον εχθρικές συνθήκες, υψώνουν το ανάστημά τους όμως και λένε ότι είμαστε αυτοί που είμαι, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε τα ίδια δικαιώματα με όλους. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. κατάσταση στην Ουγκάντα, πραγματικά είναι ανησυχητική. Ε, ο Μπράιαν έχασε τη ζωή του νωρίτερα φέτο. Πρέπει οι ε, θράστε ε, να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη. Παρενόχληση, ρητορική μίσου από τι ουγγανικέ αρχέ. Αυτά όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα. Καλούμε την κυβέρνηση τη Ουγγάντα να σεβαστεί πλήρω τα δικαιώματα τον ΛΟΑΤΚΙ. Όχι μόνο να σταματήσει η ρητορική μίσο, αλλά η νομοθεσία τη χώρας να μην κάνει διακρίση σε κανέναν λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητα. Σήμερα στηρίζουμε όλου όσου αγωνίζονται για τα δικαιώματά του στην Ουγκάντα, αλλά και παντού. Είμαστε στο πλευρό σα εμεί από την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ματία. Muito obrigada, Sr. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες γιατί υπήρξε συνένεση μεταξύ μας ε, για να δοθεί υποστήριξη από το σώμα ε, σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα να καταλάβουμε είναι πω ε, η διακριτική μεταχείριση λόγω γενετή προσανατολισμού είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Ουγγάντα. Συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, ακόμη και σε κάποια κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι πρέπει την προσοχή μα να την εστιάσουμε στην ανάγκη να προωθήσουμε την ισότητα για όλου ε, και εντό Ευρώπη και εκτό Ευρώπη. Και σε χώρε όπω η Ουγγάντα βεβαίω. πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι λέει η Συμφωνία Κοτονού. Καμία διακρίση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Είδαμε του τελευταίους μήνες ε, όμως ε, την ομή δολοφονία ενός ακτιβιστή, του Μπράιαν Βάσβα. Δεν πρέπει να δεχθούμε τέτοιες πράξεις. Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να μην υπάρχει καμία διάκριση λόγω ε, της ε, το προσανατολισμό σε κανένα μέρος του κόσμου. Η κυρία Κάρσπλο για ένα λεπτό. not be a crime. Η ομοφιλοφιλία δεν μπορεί να είναι έγκλημα και όμως χαρακτηρίζεται σαν τέτοιο σε 70 χώρες. Και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια μέλη της κυβέρνησης της Ουγγάντα ε, υποστήριξαν ε, κυρώσεις και ποινές ε, και επίσης και τη θανατική ποινή για ομοφιλοφιλικές ε, ενέργειες. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι το ποινικά κολάσιμο και οι ΛΟΑΤΒ γενικά δυστυχώς υφίστανται βία και διακρίσεις. Η κυβέρνηση όχι μόνο το επιτρέπει αλλά το τροφοδοτεί ουσιαστικά. Εάν πράγματι θέλουμε να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε να καταργήσουμε παντού τη θανατική ποινή, θα ήθελαμε να γνωρίζει η κοινότητα ΛΟΑΤ της Ουγγάντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του στηρίζει. Γιατί η αγάπη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι έγκλημα. Κυρία Γουόρτ, για ένα λεπτό. In light υπό το φως ε, της ε, αύξησης ε, των επιθέσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγάντα το σημερινό ψήφισμα έχει μεγάλη σημασία. Τρεις γκέι άνδρες και μία τρανς γυναίκα δολοφονήθηκαν φέτος. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Μπράιαν Ρουάσχα, ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ που δολοφονήθηκε στο σπίτι του η επιδείνωση των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών είναι πάρα πολύ ανησυχητική ε, συμπεριλαμβανομένης ε, και της παραβίασης των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ελευθερίας έκφρασης ε, και ισότητας των φίλων. Το ψήφισμα αυτό ζητάει να υπάρξει μια συνεργασία με την Ουγγάντα. Θα πρέπει να μην υπάρχουν τιμωρητικοί νόμοι ή πρακτική που στιγματίζει τους ανθρώπους αυτούς. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή μέσω στήριξης ε, των ΜΚΟ και εφαρμογής ε, των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών. Ζητάμε επίσης ε, να μην υπάρξει καμία διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό. Οι παλαιοί απεικιοκρατικοί νόμοι δεν έχουν θέση τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τομπέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους που συνεργάστηκαν. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη αυτού ανεξαρτήτως του σεξιαλικού τους προσανατολισμού μπορούν να είναι ελεύθεροι και ασφαλείς. Δυστυχώς στην Ουγγάντα η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή πλέον και η πρόταση η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση σχετικά με την εισαγωγή της στατατικής ποινής για τέτοιου είδους ε, πράξεις ε, είναι κάτι το καταδικαστέο. Είναι προφανές ότι απαιτείται μια ξεκάθαρη δήλωση ότι οι ναι, νέες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Η ομοφοβική και η ρητορική τους δυστυχώς ακούγονται όλο και περισσότερο έτσι οδηγούμεθα σε δολοφονίες ομοφιλόφιλων προσώπων και αυτό απάδει με τη δημοκρατία και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι και αλλιώ η αναπτυξιακή βοήθεια συνοδεύεται από προϋποθέσεις συνδεόμενες με τη σειρά τους με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν την κοινωνία των πολιτών πρέπει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση για την επιβίωση των πολιτών των χωρών αυτών. Θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε το κράτος δικαίου. Των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γουάλς. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται να χρησιμοποιείται ο σεξουαλικό προσανατολισμό για παραβιάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ουγγάντα και στην Ινδονησία είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάκριση κατά τον ΛΟΑΤΚΙ παραβιάζει τις βασικότερε αρχέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω αυτέ αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να αντιδράσει αυτέ αυτές τις παραβιάσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα δράσουν και άλλα θεσμικά όργανα. Έχει μεγάλη σημασία να ζητήσουμε από τη νέα Κομισιόν και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τι κατευθυντήριε γραμμέ περί ΛΟΑΤΚΙ, να περιλάβουν τα μέλη των κοινοτήτων αυτών στον διάλογο με τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Πρέπει να υπάρχει διάλογος για να αλλάξουν οι νόμοι διακριτικής μεταχειρίσης, να καταπολεμηθεί η ομοφοβία κατά των κοινοτήτων αυτών και να προστατεύσουμε τις ε, κοινότητε αυτές. Πρέπει να ηγηθούμε ως ε, μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και εγώ, εάν η δολοφονία τριών γκέι ανδρών και ενός ε, τρανς ε, συνέβαινε στην Ιρλανδία θα ήταν συγκλονιστικό. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Άγιος Σαλίμπα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ δυστυχώς δεν γίνονται σεβαστά ε, σε ολόκληρο τον κόσμο και μεταξύ άλλων χωρών αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε στην Ουγγάντα. Ε, Βίες επιθέσεις κατά τον ΛΟΑΤΚΙ πρέπει να έχουν το δικαίωμα ε, στην προστασία, να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους οι άνθρωποι αυτοί. Επομένως, η βία σε βάρος τους ε, ε, είναι κάτι το οποίο δείχνει μίσος προκατάληψη. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία Μόνο έτσι θα αποφευχθούν τέτοια εγκλήματα. Πρέπει να δείξουμε όλοι σθένος ε, και να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα παντού στην κοινωνία όπου τα συναντούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ ανά τον κόσμο, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τέτοιου είδους διακρίσεις και να φροντίσουμε όλοι ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ε, φύλου να έχουν το δικαίωμα να είναι ίση απέναντι στον νόμο. Η Μάλτα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για την Ευρώπη. Έχουν ψηφιστεί πολύ προοδευτικοί νόμοι και για τους γάμους μεταξύ ομόφυλων. Ε, Ομάδα Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ροντρίγκε Ράμος. Ευχαριστώ. Θυμόμαστε ακόμα τις συζητήσεις που είχαμε το 2014 όταν ε, στην ε, Ουγγάντα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο για να τιμωρείται με θανατική καταδίκη ε, η ομοφιλοφιλία και ακριβώς η πίεση της διεθνούς κοινότητας οδήγησε στην απόσταση του νόμου αυτού. Ωστόσο, η ομοφιλοφιλία στην Ουγγάντα εξακολουθεί να τιμωρείται, είναι στο ποινικό κώδικα και τιμωρείται με αυστηρές ποινές σήμερα και Καθημερινά θα έλεγα βλέπουμε πολύ δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους ε, ΛΟΑΤΚΙ, δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία ε, και πραγματικά ε, ενδεχομένως γίνει ακόμα πιο αυστηρή η νομοθεσία με πιο αυστηρές ποινές μεταξύ αυτών και η θανατική καταδίκη. Μακάρι να μην είναι έτσι. Πρέπει να στείλουμε όμω με το ψήφισμά μα ένα πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα. Ούτε ένα βήμα προ τα πίσω δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Αντίθετα, πρόοδο θέλουμε προ τον εκδημοκρατισμό στην κοινωνία. Στην Ουγγάντα μόνο βήματα προς τα εμπρός πρέπει να γίνουν. Από ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας δεν είναι έγκλημα η ομοφιλοφιλία. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον διάλογο. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων, το λόγο έχει ένα λεπτό ο κύριο αντρεσεν Άντρεσεν. Αρχέ Αρχές Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χρονο Μπράιαν Γουάσουα στην Ουγγάντα. γιατί ήταν ομοφυλόφιλος. Δέκα μαχαιριές έφαγε στο κεφάλι. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράλληλα ότι εισάγεται η θανατική ποινή για τους ομοφιλόφιλους. Ε, υπάρχει μια συνεχής ε, προπαγάνδα και ένα κυνήγι μαγισσών. Κυνήγι μαγισσών το οποίο πρέπει να τελειώσει. Και μόνο και η συζήτηση περί θανατικής ποινής βλάπτει μαζικά και πρέπει να την καταδικάσουμε. Όλοι οι άνθρωποι θα ε, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζουν και να αγαπούν ελεύθερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 578 εκατομμύρια ετησίως ε, στην Ουγγάντα. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε μια ευθύνη. Σε 70 χώρες παγκοσμίω είναι ποινικοποιημένη η ομοφιλοφιλία. Σε 9 υπάρχει θανατική ποινή. Οπότε ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώσει αυτή η πρακτική. Να είναι όλοι οι άνθρωποι ελεύθεροι παγκοσμίως. Ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Κάνκο. You have the floor. Two African uh, countries. Υπάρχουν ε, πολλές χώρες στην Αφρική οι οποίες τιμωρούν τον γενετήσιο ομοφιλοφιλικό προσανατολισμό με τη θανατική ποινή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πραγματικά όταν ήμουν νέα δεν μπορούσα να φανταστώ μια διαφορετική ζωή αν δεν ήμουν ετεροφιλόφιλη. Είναι η κατάσταση απαράδεκτη και δυστυχώς χειροτερεύει από ό,τι φαίνεται. Για να πετύχουμε λοιπόν κάποιες ε, αντιλήψεις ε, συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αρκεί να είναι κανείς θλιμμένος ε, ή να καταδικάζει αλλά να προωθεί τον διάλογο, να προωθεί τη συνένεση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ληφθούν μέτρα για την προστασία των κοινοτήτων ΛΟΑΝ. Ε, τα πολιτικά συστήματα και οι δυνάμεις καταστολής θα πρέπει να τερματίσουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Στα πλαίσια του διαλόγου που έχουμε με τις χώρες αυτές πρέπει να προωθήσουμε την αμοιβαία κατανόμη, κατανόηση και την ανοχή. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ροντρίγκες Παλό. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ουκάντα οι και σχέσεις τιμωρούνται με διαβίου κάθερξη ότι είναι παραφύση. Ε, κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν ε, από το Μεσαίωνα σαν ιδέα. Και πολλές ε, χώρες έχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Ο Υπουργό ηθικής και Ακαιρεότητα θέλει να θανατώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Παρότι το 2014 το συνταγματικό, συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε αυτέ τι προσπάθειε. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν σταυροφορία κατά του κακού κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε εμεί μαθήματα, γιατί έχουμε θρησκευτικά λόμπι που κάθονται εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο και σε άλλα εθνικά κοινοβούλια. Και χθε είχαμε συζήτηση για μια οδηγία κατά δεκτική μεταχείριση εδώ. Δέκα χρόνια όμω είναι μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο αυτή η οδηγία. Έχουμε επίση την ομοφιλοφιλική και τρανσφοβική άκρα δεξιά που είναι εδώ σε αυτά τα έδρανα. Ε, να μην τιμωρήσουμε λοιπόν την Ουγγάντα και τον ευάλωτο πληθυσμό τη ακόμη περισσότερο περισσότερο όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να λογοκρίνουμε και να καταγγέλουμε τέτοιου είδους ε, πρακτικές, αλλά να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ και όλα τα κράτη να μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο σε όσους διώκονται λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Αυτό πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε όταν ε, πρόκειται για την Ουκάντα. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ομιλητών εκ των πολιτικών ομάδων. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Μπούλ για ένα λεπτό, μη εγγεγραμμένος. Discrimination Διακρίσεις ε, επί τη βάση της, ε, του γενετήσου προσανατολισμού είναι κάτι το απαράδεκτο. Υπάρχει μισό εκατομμύριο ομοφιλόφιλων στην Ουγγάντα, παρόλα αυτά είναι παράνομοι έτσι και αλλιώς απαγορεύονται οι γάμοι μεταξύ προσώπων ε, του ιδίου φύλου και ε, καταπιέζονται κοινωνικά και υφίστανται φυσική βία. Δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει. Ήδη από το 2007 ε, το 97% πίστευε ότι πρέπει να απαγορευτεί η ομοφιλοφιλία αλλά ε, πρόσφατα έχει πέσει ο αριθμός αυτός, το ποσοστό αυτό στο 54%. Κάποιες αλλαγές δηλαδή συμβαίνουν. Λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να παρέμβουμε λοιπόν ε, σε μια δημοκρατική χώρα ε, και τα λόγια που λέμε εδώ στην ουσία δεν έχουν κανένα νόημα και δεν επηρεάζουν καθόλου τη ζωή των ομοφιλόφιλων στην Ουγγάντα η Ουγγάντα μόνη της θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να επιτρέψει στα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ να ζήσουν και να αγαπούν εν ειρήνη. Έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκονζάλες. Gracias, presidente. África nos necesita. Η, η Αφρική το χρειάζεται, η Ουγγάντα το χρειάζεται αλλά η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να συνοδεύεται από την προϋπόθεση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤ. Πρόκειται για ένα καθοριστικό στοιχείο, το περιλαμβάνει αυτό η ίδια η συνθήκη δυτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της αναγνώρισης του καθολικού χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 32 εκατομμύρια ευρώ δίδονται στην περιοχή αυτή της Αφρικής ε, της βάση. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Συμφωνία του Κοτονού λέγει ότι εάν δεν υπάρχει ο σεβασμός αυτός μπορεί να διακοπεί η χρηματοδότηση. Το κοινοβούλιο αυτό λοιπόν πρέπει να προασπίσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ χωρίς διακρίσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Μπένιον για ένα λεπτό. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ έχουν αφαιρεθεί από την σχετική νομοθεσία εδώ καιρό. Ε, ιστορικά παρενοχλείται από το κράτος ε, και την αστυνομία και τώρα έρχεται ο νόμος ε, περί θανάτωσης ε, των ε, γκέι. Δεν ποινικοποιούνται απλώς οι ίδιες οι πράξεις, αλλά και όποιος διαδίδει σχετικές πληροφορίες. Έτσι θα οδηγηθούμε σε κυνήγι μάγισσών και εξοδικαστικές εκτελέσεις ακόμα. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αφήσει να συμβεί αυτό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Ουγγάντα ότι το δικαίωμα σεξουαλικότητα και την έκφρασή της και η ελευθερία από διακρίσεις βασίζεται στα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και, από, και στο διεθνές ανθρωπιστικό δικαίωμα. Επιπλέον, σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η Ουγγάντα έχει σχετικές υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από πέντε χρόνια πολύ ε, ανακουφιστήκαμε όταν η Ουγκάντα απέσυρε την ε, θανατική ποινή. Αλλά τώρα έχουμε ένα νέο νόμο ο οποίος ε, προτείνεται. Η αναπτυξιακή βοήθεια στην Ουγκάντα μεταξύ του 2014 και 2020 ανέρχεται σε 578 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά. Αλλά τα λεφτά αυτά είναι υπό όρους. Υπάρχουν σαφείς ε, δηλώσεις στην συμφωνία ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό εμείς οι πράσινοι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετηθεί σαφώς κατά αυτών των εξελίξεων στην Ουγκάντα. Έχουμε διάβρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντέλη. Thank you, President. I am of course... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω είμαι κατά τη ανατική ποινή. Τελεία. Αλλά το γεγονό ότι το σκέφτονταν για ερωτικά εγκλήματα είναι απαράδεκτο. Αλλά ας είμαστε σαφεί. η ποινικοποίηση τη ομοφιλοφιλίας υπό οποιαδήποτε μορφή νομοποιεί το ομοφοβικό μίσος και αποτελεί θανατική ποινή για πολλούς ανθρώπους. Και βεβαίως ε, είμαι πλήρως αλληλέγγυα με τα θύματα στην Ουγκάντα και τους ακτιβιστές στην περιοχή αυτή. Αλλά είναι περίεργο ότι κάποιοι εδώ μέσα θέλουν να προσθέσουν σε αυτό το ψήφισμα και ε, συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και είμαστε κάποιος φάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Ουγγάντα για να βρούμε διακρίσεις ε, κατά τον ε, ΛΟΑΤΚΙ. Για πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη η αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά τις δεξιές προκαταλήψεις και τομήσεις υπάρχει στα δικά μας τα κράτη. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα δικά μας πρώτα. Το, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Thank you. Ευχαριστώ. Ήδη είναι ταπεινωτικό ε, το να μην μπορεί να παντρευτώ τον άντρα τον οποίο αγαπώ ε, σε όλες τις 28 ε, χώρες. Θα έπρεπε να έχω αυτό το δικαίωμα, αλλά τουλάχιστον γνωρίζω ότι δεν απειλεί τη ζωή μου όταν περπατώ χέρι-χέρι ε, με τον ε, συντροφό μου, στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον της Ευρώπης. Ε, εδώ βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα και θάματα στην Ουγγάντα. Σε μόλε κόντο, υποτιθέμενος υπουργό ηθικής και καιρότητα, πρέπει να ντρέπεται. Τι κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις αδυναμίες της κυβέρνησης. Χρησιμοποιεί ως αποδοπομπείο τράγω την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ σε όλες τις χώρες και στην ε, ε, Ουγγάντα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους πούμε ότι δεν είστε εσείς το πρόγραμμα, πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι κυβερνήσεις σας που αποτυγχάνουν, σας χρησιμοποιούν ως εξυλαστήρια θύματα. Πρέπει να σταθείτε ισχυροί, έχετε την αλληλεγγύη μας, την ε, υποστήριξή μας. Ο αγώνας που δίνεται δεν γίνεται μόνο στην Αφρική, στην Ασία, γίνεται παντού και εμείς είμαστε στο πλευρό σας σε αυτή τη μάχη που δίνεται και πρέπει να απακυρωθούν όλοι αυτοί οι απεικιοκρατικοί νόμοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί έξι αιτήματα. Τα κάνω και τα έξι αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριο Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες του ψηφίσματος, καθώς και όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Γιατί μιλάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια φωνή αρνούμαστε να δεχτούμε αυτή την πολιτική πραγματικότητα με αυτό το νομοσχέδιο στην Ουγγάντα, το σκανδαλώδες αυτό νομοσχέδιο. Εσείς, Επίτροπε, ή ο προσεχής, ο επόμενος που θα αναλάβει καθήκοντα, έχετε την ευθύνη. Δεν πρέπει να στέλνουμε χρήματα σε χώρες ε, που παρενοχλούνται και ε, ε, αντιμετωπίζονται, διώκονται ουσιαστικά οι κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ. Πρέπει η βοήθεια που στέλνουμε στην Ουγγάντα να στέλνεται και ξέρουμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για σήματα ποσά. Με τα λόγω γνώσεως μπορούμε να στέλνουμε χρήματα σε χώρα που καταδικάζει θάνατο τους ομοφιλόφιλους. Αυτά είναι σκανδαλώδη πράγματα. Δεν μπορούμε να στέλνουμε χρήματα σε μια τέτοια χώρα. Το ψήφισμα αυτό πρέπει να ε, δώσει όθηση στην Κομισιόν να αλλάξει την πολιτική Για ένα λεπτό, κύριος Λόπες Αγγιλάρα. Επίτροπε Μίμητσα, Πρόεδρε, Είχαμε συζητήσει λοιπόν τα θέματα αυτά στο Στρασβούργο, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσοι είμαστε παρόντες έχουμε ε, πραγματικά είμαστε πεπισμένοι εναντίον κάθε μορφής ε, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εναντίον της θανατικής ποινής ε, και εδώ σε αυτήν την προφανή περίπτωση ποινικοποίηση της σεξουαλικής ομοφιλοφιλικής δραστηριότητας θα έλεγα ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, πράγματι ένα μεγάλο ε, κομμάτι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει στη βοήθεια για την ανάπτυξη και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτά δεν είναι προφανώς συμβατά με μέτρα αυτά που παρεμποδίζουν τον έρωτα μεταξύ των ανθρώπων. Είναι λοιπόν απαράδεκ, ότι είναι ασύμβατες οι δραστηριότητες αυτές και οι χώρες αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από τις σημαντικές πιστώσεις οι οποίες τρέφονται μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις χώρες. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Thank you. I'd like to ask Ευχαριστώ. Μια ερώτηση όχι μόνο στους συναδέλφους και σε όλους που μας ακούν. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να ζει κανείς, να εργάζεται, να αγαπά ε, και ποια είναι η κυβέρνηση, ποια είναι η ιδεολογία, ποια είναι η θρησκεία που θα σου αφαιρέσει αυτό το ε, ανθρώπινο δικαίωμα. Με την ψηφοφορία αυτή λοιπόν σήμερα και με την προσπάθειά μας σαν ακτιβιστές και σαν βουλευτής στην χώρα μου ε, μπορώ να πω ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα ε, να ακυρώσει την αξιοπρέπεια των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΒΟ ούτε στην Ουγγάντα ούτε πουθενά άλλο. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να κάνουμε την προσπάθεια αυτή να καταπολεμήσουμε την κατάσταση και στην Ουγγάντα και στην Ευρώπη. Για ένα λεπτό κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ε, ως προς τότε φυσικά ομές, επιθέσεις ε, σε ανθρώπους που απλά είναι διαφορετικοί είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο. Απολύτως απαράδεκτη είναι και η ε, προσέγγιση και η ε, πολιτική της κυβέρνησης της Ουγκάντας που θέλει να εισαγάγει μέχρι και τη θανατική ποινή για ανθρώπους που απλά είναι διαφορετικοί είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι ένα βήμα πίσω στο μεσαίωνα. Και η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Πρέπει οι θέσεις μας να γίνονται ε, αισθητέ μέσω των πολιτικών μας και μέσω της βοήθειας που δίνουμε ή δεν δίνουμε με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη δεκαετία του 60 στην Τσεχία η ομοφιλοφιλία ήταν παράνομη. Αλλά άλλαξαν τα πράγματα. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί στην Γκάντα. Λόγο έχει για ένα λεπτό ο Τσιχοντάρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το πρόβλημα του 21ου αιώνα είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλιώ ε, δεν θα υπάρχει ζωή. Κάποιες χώρες επιστρέφουν στον ε, μεσαίωνα και θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην ελεύθερη έκφραση ε, παραβιάζονται όπως στο μεσαίωνα. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να βρουν κοινά μέτρα και σαφή κριτήρια έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μην συμβαίνουν στο μέλλον. Και πρέπει να έχουμε μια κοινή αντίληψη όταν παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί καμιά φορά είναι δύσκολο να δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα εντός ε, και εκτός. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Κομισιόν να φροντίσουν ε, να είμαστε στον 21ο αιώνα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μάξοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερω που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρτήσει ένα πολύ ισχυρό ψήφισμα κατά τη θέσπιση αυτή τη νομοθεσία ε, ε, που ουσιαστικά προβλέπει και θανατική ποινή ε, για διάφορε περιπτώσει σεξουαλικού προσανατολισμού. Το μπαλάκι τώρα είναι στο γήπεδο τη Κομισιόν και πρέπει να ακολουθήσει ε, την προσέγγιση που τις συνιστούν οι προλαλήσαντες. Ομοφιλοφιλία δεν είναι ούτε σφαγή, ούτε κλοπή, ούτε οτιδήποτε. Ο ε, λιθοβολισμός μέχρι θανάτου, η θέσπιση εκ νέου της θανατικής ποινή για τέτοιου είδους εντό αγωγικών αδικήματα είναι κάτι απαράδεκτο. Πρέπει να ψώσουμε τη φωνή μας σε βάρος τέτοιου είδους διακριτικής μεταχείρισης και ελπίζω και χαίρομαι ε, να στείλουμε ένα μήνυμα από πλευράς Κοινοβουλίου στην κοινότητα των ΛΑΤΚΙ στην Ουγγάντα. Είμαστε στο πλευρό του και δεν μπορεί κανεί να του τιμωρεί μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν όπω γεννήθηκαν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙΑΙ. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, το λόγο έχει ο Επίτροπο κ. Μίμητσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ότι οι ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγάντα επί σειρά ετών αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία, μεταξύ των οποίων και εγκλήματα μίσους. Τα τελευταία σχόλια του Υπουργού της χώρας ε, περί της πιθανότητας να προταθεί νέος νόμος κατά της ομοφιλοφιλίας στο Κοινοβούλιο που πιθανώς ε, θα προβλέπει και τη θανατική ποινή είναι ένα θλιβερό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας η άμεση επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης και της Προεδρίας που διαβιβάστηκαν και μέσω διπλωματικών διάβλων στους πρέσβεις ε, των κρατών μελών ε, ε, επιβεβαίωσαν ότι δεν συντάσσεται τέτοιος νόμος. Άρα πρέπει να θεωρήσουμε αυτό το σχόλιο πολύ ανησυχητικό αλλά δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι μια τέτοια δημόσια δήλωση από έναν υψηλό βαθμό υπουργό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λυπηρε αντιδράσεις και περαιτέρω διακρίσεις ή και βία κατά τον ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ειδικά νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα, έτσι ώστε η σεξουαλική ταυτότητα και προσανατολισμός ε, υπό ε, οποιασδήποτε συνθήκες να μην ε, τιμωρούνται ποινικά, ειδικά ε, μέσω της εκτέλεσης, καθώ καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της ανατικής ποινής υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Η διακριτική αυτή μεταχείριση παραβιάζει τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας διαβεβαιώ πως όλες μας οι υπηρεσίες και ειδικά η αντιπροσωπεία μας στην Καμπάλα παρακολουθούν την κατάσταση στενά και θα μεταφέρουν τα μηνύματά μας ε, και την δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κατάλληλο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Η επόμενη συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αφορά την Αίγυπτο. Πριν από την έναρξη συζήτηση θα ήθελα και πάλι να σας ενημερώσω ότι για να ζητήσετε το λόγο με τη διαδικασια the Eye ή για να θέσετε ερώτηση με γαλάζια κάρτα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τον συνήθι τρόπο εγγραφής και το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής. Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να έχετε μαζί σας πάντα την κάρτα πληροφορίας. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε για τη διαδικασία Catch the Eye, σας παρακαλώ μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα χωρίς να περιμένετε το τέλος της συζήτησης. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο εκ των η εκ των συντακτών κυρία Νόημαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Σεπτέμβριο χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους στην Αίγυπτο και το ίδιο ε, έγινε σε πάρα πολλές πόλεις, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, κατά της διαφθοράς ε, και κατά της ε, υπεξαίρεσης πόρων που υποτίθεται θα πήγαιναν για την οδοποιία και άλλα έργα υποδομόνα. 4.300 άτομα έχουν μπει φυλακή και εκατοντάδες παιδιά μεταξύ αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και τα κοινωνικά μέσα και γενικά ε, ο τύπος ε, επιτηρείται είναι ξεκάθαρος. Εσύ δεν δέχεται καμία κριτική ε, και καταστέλει την κριτική. Σήμερα πολλοί κόσμος μπορεί να μιλήσει μόνο αν μάλλον με τον κίνδυνο να, να πρέπει να εξοριστεί ή να μπει φυλακή. Ε, βλέπουμε επίσης εξαγωγή τεχνολογίας και όπλων ε, προς τη χώρα. Ήμουν εισηγήτρια ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν εύκολη η συζήτηση για αυτό το ψήφισμα, διότι πραγματικά είναι σημαντικό να συναγάγουμε τα συμπεράσματά μας. Ευτυχώς παρά τις διαφωνίες μας όλοι οι εισηγητές συμφωνήσαμε και είμαι περήφανη γι' αυτό, διότι ναι μεν συμφωνούμε ότι είναι ένας εταίρος της Ένωσης η Αίγυπτος, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι πλέον πλέον του καθεστώτο. Πλωμένω πρέπει να πάψουμε το business as usual με τον Σίση. Θέλουμε ελευθερία για αυτού που διαδηλώνουν και συγκεκριμένα δεν θέλουμε κατασκοπία να ε, επιτρέπεται να κερδίζουν κάποια χρήματα στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να στείλουμε λευκό επιταγές πλέον ε, στη χώρα. Θέλουμε όμως τα χρήματα μας να πηγαίνουν στην ενίσχυση κοινωνία των πολιτών. Και στρέφομαι στην Κομισιόν. Επιτέλους ε, ξεκάθαρες δηλώσεις διπλωματικού χαρακτήρα κτλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το μυαλό μου είναι στραμμένο στην Αίγυπτο και όταν έχουμε υπόψη μας πόσοι άνθρωποι περιμένουν ε, όταν καταπατώνται τα δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Ελπίζω με αυτό το ψήφισμα σήμερα να δώσουμε ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Ούρμπαν Κρέσπο. Ευχαριστώ. Για μια ακόμη φορά, αγαπητέ πρόεδρε, μιλάμε για την Αίγυπτο. Για ποιο λόγο? Λόγω της ομής καταστολής ε, κατά των ε, κοινωνικών κινητοποίησεων. Όλες οι συναντιόταν στα Ηνωμένα Έθνη με τους ηθήνοντες από όλο τον κόσμο. Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι φυλακίζονταν. Έχουμε ανθρώπους που αγνοούνται, άλλους που έχουν βασανιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει απ' την άλλη. Ενώ τα κράτη-μέλη πουλάνε στρατιωτικό εξοπλισμό που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ε, στη χώρα για να καταστέλουν ε, το Αιγυπτιακό λαϊκό κίνημα. Δεν προστατεύει λοιπόν στην Αίγυπτο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε καν ζητάμε κάτι τέτοιο. Λέμε απλά ότι δεν μπορεί να καλύπτει ε, την ε, δικτατορία ε, στη χώρα αυτή η Ένωση. Απαιτούμε την δημοσιονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο προς την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Ζητούμε αναστολή των συνομιλιών για εμπορική συμφωνία με την Αίγυπτο μέχρι να σεβαστεί η χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε πραγματικό εμπάργκο στα όπλα και Θέλουμε συνεργασία σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Τέλος, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε μέτρα, όχι συνεργασία με τη δικτατορία. Για να μην είναι καινογράμμα τα λόγια που λέμε. Για να μην ξαναμιλήσουμε στην Ολομέλη για την Αίγυπτο. Τέλος, να ληφθούν μέτρα και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Οστρεβίτσιου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο έδειξαν πόσο λίγος είναι ο χώρος για την ελευθερία έκφρασης και ε, το ειρηνικό συνέρχεσθε στη χώρα. Βλέπουμε δυστυχώς δυσανάλογη χρήση βίας σε βάρος διαδηλωτών, παράνομη συμπεριφορά απέναντι στους υπέρασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορισμό της δραστηριότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αυτό που με ανησυχεί όμως περισσότερο είναι το γεγονός ότι η ηγεσία της Αιγύπτου ε, χρησιμοποιεί και περισσότερο την καταπολέμηση της δημοκρατίας ε, ως μέσο στηρικής πολιτικής για να φημώσει τους πολιτικούς της ε, αντιπάλους και να σταματήσει τη δημόσια κριτική ο διάλογος μεταξύ της ηγεσία της χώρας και της κοινωνίας της Αιγύπτου είναι δυνατόν να γίνει μόνο εάν ανταποκριθεί η ηγεσία στις προσδοκίες των πολιτών και κάνει τις τόσο σημαντικές και απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να σε διάφορου τομείς. Εμεί πρέπει από την πλευρά της Ένωσης ε, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και με χρηματοοικονομική υποστήριξη των περασπιστών ε, της, ε, και της κοινωνία των πολιτών. Έχει η κυρία Αρένα για 1,5 λεπτό. Ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου οι αντικυβερνητικοί έχουν διαδηλώσει στο σύνολο της Αιγύπτου σε όλες τις πόλεις άνω των 4.000 αυθαίρετων συλλήψεων, δημοσιογράφων, δικηγόρων, προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι φυλακισμένοι με βαριές κατηγορίες και με κατηγορίες τρομοκρατίας δεν έχουν επαφή με τους δικηγόρους τους, δεν έχουν επαφή με τις οικογένειές τους, πολλοί βασανίζονται, δεν τους παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες, ένα πλαίσιο καταστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, το δικαίωμα του συνέρχεστε όπως και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέσω πρόσωπα εδώ. Νταμισάντ, Μπελχαντά, Ντεχαλτά, Αμπές και χιλιάδες άλλοι που είναι πια φυλακισμένοι. Καταδικάζουμε τις δράσεις της κυβέρνησης του Καΐρου και ζητάμε την Αίγυπτο να ολοκληρώσει τη μετάβαση στη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευματίσει την οικονομική βοήθεια αν δεν ολοκληρωθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πάβουν να εξάγουν όπλα που χρησιμοποιούνται εις βάρος των ανθρώπων. για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους αδελφούς στο ψήφισμα αυτό. Ζητάει από την Αίγυπτο να ανοίξει στον κόσμο. Η κριτική που ακούσαμε κατά των ηγετών της ε, Αιγύπτου είναι επικοδομητική κριτική αναφέρεται σε σημαντικά πράγματα ε, τα οποία είναι στραβά στην Αίγυπτο έχουμε κάνει καλή δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλη μας η βοήθεια πήγε στα χέρια τρομοκρατών. Τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτίζουν νοσοκομεία και βελτιώνουν την κατάσταση υγείας. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας ανοιχτός διάλογος με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Αίγυπτος δεν συμμορφώνεται με τις ε, διεθνείς ε, απαιτήσεις ε, και προδιαγραφές, παραδείγματος χάρη για την δίκαιη δίκη η νομική προστασία των ε, αδυνάμων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά και οι διάφοροι άνθρωποι απλά εξαφανίζονται. Θέλουμε λοιπόν η Αίγυπτος να μας δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μας. Πρέπει επίσης να αναζητήσουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες που εξαφανίστηκαν στην Αίγυπτο και δεν έχουμε ακούσει τίποτα, καμία εξήγηση από την Αίγυπτο. Ναι, να αλλάξει η πολιτική μας ε, απέναντι στην Αίγυπτο. Πράγματι πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ ε, αυστηροί σε κάποιους ε, τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στο θέμα του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Λαϊκού Κόμματο, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριο Κέλλη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε συζητήσει ξανά το ίδιο θέμα Ενθυμίστε γενικά και το ψήφισμα που είχαμε περάσει πριν από αρκετό καιρό. Ενθυμούμεθα την υπόθεση ενός νέου ανθρώπου που είχε φυλακιστεί στην Αίγυπτο, δεν είχε περάσει από δικαστήριο, δεν του είχε δώσει καμία, δεν του είχαν δώσει καμία δυνατότητα να αμυνθεί αλλά μετά από τις παρεμβάσεις μας και μετά από τις πιέσεις μας απελευθερώθηκε και έχει επιστρέψει τώρα στην Ιρλανδία και δεν δημιουργεί βέβαια κανένα θέμα για την Αιγυπτιακή κυβέρνηση αυτό. Δυστυχώς 4.300 είναι αυτοί που συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Κάποιοι από αυτούς έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον ίχνη τους. Και πάνω από 100 ε, νέοι, ανήλικοι μάλλον, είναι πια στη φυλακή. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε την ίδια πίεση για μια ακόμη φορά προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, να μας ακούσουν και να απελευθερώσουν τους πολίτες αυτούς. Κατανοώ βέβαια ότι η Αίγυπτος έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα α, της α, τρομοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα σαν χριστιανός θα έλεγα, και σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απαιτείται να διασφαλίσουμε ε, την υποστήριξή μας προς τους χριστιανούς της χώρας αυτής. Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είχαμε την δυνατότητα να δούμε τις εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Αίγυπτο λόγω της καταστολής, της διαφθοράς και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυθαίρετες συλλήψεις 4.000 για ειρηνική διαμαρτυρία. Δυστυχώς έτσι δράει η κυβέρνηση η Αιγυπτιακή με την καταπίεση, με την καταστολή με τον εκφοβισμό, με τις αυθαίρετες συλλήψεις και με τα στρατιωτικά δικαστήρια. Και έχουν υπάρξει φυσικά και πάρα πολλοί που έχουν ε, αυτή τη στιγμή που αγνοούνται και υπάρχουν και πάρα πολλοί ανήλικοι. Η παραβίαση λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά για τη δημοκρατία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να αλλάξει η κατάσταση στην Αίγυπτο και να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν το 2013. Όχι όπλα και τεχνολογικός εξοπλισμός για εσωτερική καταστολή και... The New Europe, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Φονδίζε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω μία περίπτωση, την περίπτωση του Ιμπραήμ Εζ Ελντίν, υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ερευνητή που ειδικεύεται στα δικαιώματα στέγασης στην Αιγυπτιακή Επιτροπή για τα Δικαιώματα και την Ελευθερία. Συνελήφθη τον Ιούνιο κοντά στο σπίτι του στο Κάιρο και απήχθη προς άγνωστη κατεύθυνση. Έκτοτε δεν είχε καμία επαφή με την οικογένειά του. Το αστυνομικό τμήμα αρνείται ότι είχε κρατηθεί ποτέ εκεί και ο Υπουργό Δικαιοσύνη δεν έχει απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα. Η σύλληψη του Ιμπραήμ ε, θεωρείται ότι σχετίζεται με την κριτική που άσκησε στην ε, κυβέρνηση τη στεγαστική της ε, πολιτικής. Είναι το πέμπτο μέλος της οργάνωσης αυτής που συνελήφθη από το 2016. Πρόκειται για μια καταστολή των υπερασπιστών ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Ζητάω από, την, ε, από το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει αυτή την περίπτωση και τις άλλες κατεπίγουσες περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση του Ιμπραήμ και των άλλων υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για την ομάδα των Πρασίνων για ένα λεπτό ο Σατούρη. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλο το θάρρος αυτών που πρασπίζονται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. 60.000 πολιτικοί κρατούμενο στην Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα εφιάλτης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έβλεπε άλλα πράγματα προσπαθούσε να έχει στη διάθεσή της δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να τα δώσει στην Αίγυπτο πριν το τέλος του χρόνου. Άμεση βοήθεια προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς συνθήκες Δυστυχώς πρόκειται για μια άμεση επίθεση ε, εις βάρος ε, των, ε, της γαλλικής κυβέρνησης η οποία πολύ όπλα στην Αίγυπτο παραβιάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Κυρία Μογκερίνη, η σιωπή σας σας καθιστά συνένοχη. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που κάνει δεν έχει παρουσία στην διεθνή σκηνή. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε μόνο την κοινωνία των πολιτών, να επιλέξουμε στοχευμένες κυρώσεις και κυρίως να σεβαστούμε το εμπάργο για τα όπλα. Και λόγο έχει Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν αναφερόμαστε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τέσσερα χρόνια μετά από την εξαφάνιση του Τζούλιο Ρετζένι, του νεαρού ερευνητή, οι Αιγυπτιακές αρχές δεν μας έχουν πει την αλήθεια για τον θάνατό του και δεν έχουν δώσει τα αποτελέσματα των διεθνών ενεργειών και των ετοιμάτων γενικά των διεθνών οργανισμών μεταξύ του οποίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Αρχών του 2018. Το να παρέχεται και να χορηγείται η δικαιοσύνη είναι καθήκον κάθε καθεστώτος και γι' αυτό θα πρέπει για τον Τζούλιο Ρετζένη να δούμε αν κάναμε τα πάντα, αν κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε. Ε, είμαστε η βασική πηγή εξωτερικών επενδύσεων για την Αίγυπτο. Η βοήθεια προς την Αίγυπτο φτάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 17-20. Η Αίγυπτος πράγματι είναι ένα σημαντικό συνομιλητής, είναι μια σημαντική χώρα για την σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και λόγω ε, ε, των συνόρων της ε, που καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο τους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Η ασφάλεια είναι παράλληλη με την διασφάλιση της αξιοπρέπειας και το κράτος δικαίου η καταστολή, η ένταση και η διεθνής κριτική μπορούν να αποσταθεροποιήσουν βέβαια την Αίγυπτο και ως εκ τούτου το σύνολο της Βορείου Αφρικής και να εμπλέξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με καταστροφικό τρόπο. Η, η αποκατάσταση της επαφής ανάμεσα στην εισαγγελία του Καΐρου και την εισαγγελία της Ρώμης πρέπει να ενθαρρυνθεί επί τη βάση της αρχής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο έτσι ώστε να οδηγηθούμε επιτέλους στην αλήθεια για τον φρικτό θάνατο του νεαρού Ιταλού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ε, να υποστηρίξει κανείς ε, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και ζητώ πράγματι να υπάρχει απόλυτο σεβασμός όλων των θρησκειών και των χριστιανών στην περιοχή και να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές για την ανακάλυψη των δολοφόνων του Ρετζένι. Δυστυχώς όμως δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζω την έλλειψη ικανοποίηση για το μανιχαϊκό τρόπο με τον οποίο εκφράζεται αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Είναι μία μέθοδος η οποία στην ουσία δαιμονοποιεί ένα συγκεκριμένο εχθρό και επιλέγει την υπεραπλουστευμένη λύση σε περίπλοκα προβλήματα. Γι' αυτό η πρόταση της κυρίας Φωτίγκα είναι μια εξαιρετική και ισορροπημένη πρόταση. Μια πλήρης καταδίκη του καθεστώτος Σίση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απομονώσει την χώρα αυτό και στην οικονομική ε, ζώνη και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσοι ακτιβιστές, πόσοι δημοσιογράφοι, πόσοι φοιτητές, ε, ΜΚΟ, γυναίκες, ε, έχουν εξαφανιστεί. Ε, πρόκειται για μια καταστολή οποιασδήποτε κριτικής ε, και βεβαίως υπάρχει και η θανατική ποινή και τόσοι περιμένουν ε, να εκτελεστούν. Βεβαίως η Αίγυπτος λέμε ότι είναι ένα σημαντικός εταίρος σε μια ανήσυχη γειτονιά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας. Ε, πράγματι πρέπει να καταπολεμηθεί ο εξτρεμισμός, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα μαζικές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυσμιστικές ε, εκστρατείες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζούλιο Ρετζένη, η οποία έχει καταλήξει σε ένα τείχος σιωπής, μια περίπτωση η οποία σωστά στιγματίζεται από το ψήφισμα αυτό. Θα πρέπει να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων πραγματικά και να παγώσουν οι σχέσεις. Αυτά θα πρέπει να γίνουν για να είμαστε σωστοί και για να αποκαταστεί η αλήθεια για τον Τζούλιο Ρετζένι. Εγώ έχει ο Μπενιφέ για Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πάλι καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο που δεν ε, μειώνουν από ό,τι φαίνεται τα βασανιστήρια και την ε, καταστολή. Δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε στενή συνεργασία με χώρες οι οποίες δεν σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες μας ή δεν βοηθούν στις δικαστικές έρευνες που αφορούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση Τζούλιο Ρετζένη. Εδώ και τρία χρόνια εκκρεμεί αυτή η υπόθεση. Η Ιταλία δεν ε, σταματάει να αναζητά την αλήθεια λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστούμε ή να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικρατεί μια, ένα κλίμα ατιμορρησίας και οι Αιγυπτιακές αρχές αρνούνται να δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τις Ιταλικές ε, αρχές. Και δεν εκδίδονται στην Ιταλία οι πέντε ύποπτοι για την υπόθεση αυτή όπως έχει ζητήσει η Αγγελία της Ρώμης. Περνάμε λοιπόν τώρα ε, στον επόμενο μιλητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2011 ήταν η ιστορική καμπή στην ιστορία της Αιγύπτου. Εκατομμύρια Αιγύπτιοι κατέβηκαν στους δρόμους με την ελπίδα για περισσότερη ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλύτερη οικονομική κατάσταση. Μετά από 8 χρόνια όμως, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία του τύπου, αυτά επιδεινώθηκαν. Ε, πίεση και ε, καταστολή χειρότερα τώρα από ότι κάτω από τον Μουμπάρακ. Η Amnesty International αναφέρει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συστηματικά βασανιστήρια και άλλες μορφές ε, κακοποίησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι απαράδεκτο. Ως απάντηση στις ε, τελευταίες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, 4.300 άνθρωποι φυλακίστηκαν αυθέρατα. Πολλοί βρίσκονται ακόμα στη φυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για βασανιστήρια. Οι ακτιβιστές μπαίνουν στο στόχαστρο και κάποια απλά εξαφανίζονται. Τα θεμελιώδη δικαιώματα καταπατούνται. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς. Έχει έρθει η χρονική στιγμή ε, να ε, βοηθήσουμε το λαό. Αυτό πλέον είναι το καθήκον μας και οφείλουμε να ε, δραστηριοποιηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπίλαν Άνταμ. Ευχαριστώ πολύ. Η Αίγυπτος είναι χώρα κλειδί για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και της ε, Βόρειας Αφρικής. Είναι ε, πολύ σημαντικός οικονομικός ε, εταίρος για την Ευρώπη και διαδραματίζει και πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η Αίγυπτος δέχεται πολλούς μετανάστες από τη Συρία και είναι επίσης και καθοριστικός εταίρος ε, στον αγώνα μας ε, κατά της τρομοκρατίας. Οι Αιγυπτιακές αρχές πολεμούν κατά των τρομοκρατών στην Χερσόνησο του Σινά. Πρόσφατα πάρα πολλοί κατέβηκαν στους δρόμους, διαδήλωσαν ε, και η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Ανάμεσα στους ε, διαδηλωτές είδαμε και πάρα πολλούς ε, οι οποίοι έχουν σχέση με τους ε, αδελφούς μουσουλμάνους ή και με το ISIS. Χαίρομαι που ο κύριος ο πρόεδρος της Αιγύπτου καταβάλει προσπάθειες για να προστατεύσει τους χριστιανούς της Αιγύπτου. Δεν τα καταφέρνει πάντα πολύ καλά. Πολλοί πέθαναν φέτος και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Χαμπίπ. Κύριε Χαμπίπ, ε, κυρίες και κύριοι, όταν ο πρόεδρος Σίση ε, Έγινε πρόεδρος της Αιγύπτου το 2014 σε ένα βασικό συμβόλαιο με το λαό της Αιγύπτου, δηλαδή η ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία για σχεδόν, με αντάλλαγμα όμως σχεδόν απόλυτο έλεγχο. Ήταν πολύ παρόμοιο ε, το συμβόλαιο με το συμβόλαιο που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η σύμβαση αυτή είναι καλή, αλλά από τη στιγμή που η σταθερότητα, η ασφάλεια και η οικονομική ευημερία συνεχίζονται. Όμως, Όταν η οικονομία σταμάτησε να αναπτύσσεται, η απάντησή του ήταν να σφίξει τα σχοινιά ε, στην εξουσία, δηλαδή να περιορίσει τις ελευθερίες των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το ίδιο ακριβώς. Εδώ, εδώ μια προειδοποίηση. Μην σφίγετε τα λουριά άλλο. Εμείς είμαστε πολύ μακριά από την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα ε, πηγαίνουμε σταθερά προς τα εκεί. Χαλαρώστε λίγο τα πράγματα α η κυρία Γκίλνη να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόσθετα. Και πάλι σηκώνομαι εδώ για να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Ο κύριο Ίσης υποσχέθηκε σταθερότητα, ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία. Δεν ε, κατάφερε τίποτα από αυτά. Το μόνο που έχει κάνει είναι να περιορίσει τι ελευθερίε ε, των πολιτών και τη κοινωνία των πολιτών. Ο Τραμπ μπορεί να συμφωνεί με αυτά που γίνονται στην Αίγυπτο. 4.300 άνθρωποι ε, συλλήφθηκαν από την έναρξη των διαμαρτυριών το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Γι' αυτό και ζητώ άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση όλων των κρατούμενων, ειδικά του Μουχάμετ Μάσρη. Ε, τι ε, απαντήσεις έχετε εσείς. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην υπόθεση του Ζούλια Ρεζίμι, ενός ε, φοιτητή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ που αγνοείται η τύχη του στο Κάιρο. Δέκα μετά βρέθη το ισορός του κάπου και φαίνεται να υπέφερε από φρικτά βασανιστήρια. Δεν έχουμε όμως καμία απάντηση έκτοτε. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει. Καμία απάντηση από τον Σίση και την κυβέρνησή του. Τι κάνουν τα εκατομμύρια που τους στέλνουμε στην Αίγυπτο σύμφωνα με την, ε, ε, ε, την πολιτική γυτνίασης. Θέλουμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία συνάδελφα. Κύριε Τσανέτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η αποσταθεροποίηση της Αιγύπτου ε, σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που θα έρθουν προς την Ευρώπη, ίσως και εκατομμύρια. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν να μην εγκλειστούν σε φυλακή. Ε, πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Μην ξεχνάμε ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι και οι Ισλαμιστές οι ακραίε λαμιστέ είναι εκείνοι που οργάνωσαν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ε, διαμαρτυρίες. Ε, γιατί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι απλά τροφή για τα κανόνια που μπορούν να τους ε, χρησιμοποιήσουν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των χριστιανών στην Αίγυπτο. Συγγνώμη, ένα μισή λεπτό έχω δικαίωμα να μιλήσω. Λοιπόν, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Αιγυπτική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, αλλά οι αδελφοί μας δέχονται, εξακολουθούν να δέχονται επιθέσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, αρχές Αιγύπτου να προστατεύσουν τους κόπτες χριστιανούς. Γιατί αυτοί αποτελούν στοιχείο σταθερότητας ε, στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε. Και συγγνώμη κιόλας που ήθελα να σας αφαιρέσω το λόγο. Πάμε τώρα στη διαδικασία ε, Catch the Eye. Πέντε έχουν ε, ζητήσει το λόγο. Πέντε συνάδελφοι. Κύριος Γεσέ Πόσπεσίτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να στηρίξω το ψήφισμα και συμφωνώ με τους συναδέρφους που έχουν επικρίνει τις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Το καθεστώς τι μας δείχνει τώρα, μας δείχνει τόσες δυσκολίες. Η Αίγυπτος φυσικά και είναι σημαντικός εταίρος, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια όταν βλέπουμε ότι καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλη μου τη ζωή ασχολιόμουν με τέτοια θέματα και ως υπουργό Δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θανατική ποινή, είναι κάτι στο οποίο γίνεται κατάχρηση τελικά. 3.000 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί χωρίς δίκη. Οι άνθρωποι αυτοί καταδικάστηκαν και νέοι και γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί στην Αίγυπτο. Είναι μοναδική περίπτωση αυτή. Πολλά δείχνει όμως αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Ο κύριος Διοντούρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Ονομάζομαι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ορισμένοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα και προκειμένου άλλοι να μπορούν να θριαμβεύουν. Και τελικά τι γίνεται, βάζουμε ε, τα όρια ανάμεσα στη δημοκρατία και την δικτατορία. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μιλήσει κατά το παρελθόν για ένα σωρό πράγματα, για ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάσει κτλ. Γράφει ωραία κείμενα, αλλά δεν έρχονται συγκεκριμένα μέτρα. Δεν κάνει τελικά τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν έχω να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Κάνω έκκληση προ την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φυλακισμένοι βρίσκονται στη φυλακή βάσει πολιτικών κριτηρίων. Αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να σταματήσει και να απελευθερωθούν. Ευχαριστώ η κυρία Ντέλη Κλακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει μια θλιβερή ηρωνία στο ψήφισμα αυτό. Γιατί πρόκειται για copy-paste ουσιαστικά του ψηφίσματος που πέρασε πριν από ένα χρόνο. Και όμως η κατάσταση επιτόπου στην Αίγυπτο επιδεινώνεται. Και εγώ βρίσκω ότι χρησιμοποιούμε διπλό λόγο εδώ στην Ευρώπη, γιατί για να προχωρήσουμε πρέπει να κοιτάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Και ναι, μεν το ψήφισμα εκφράζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιθυμίες του Αιγυπτιακού λαού να έχει ελευθερία, ευημερία και μια δημοκρατική κοινωνία. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχάρει τον Σίση, τον πρόεδρο Σίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ε, πρόεδρος ε, συνελήφθη και ήταν από, στην απομόνωση και τελικά πέθανε ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος. Οπότε λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε, να έχουμε υπόψη μας με ποιους συνεργαζόμαστε, όπως για παράδειγμα είναι η Σαουδική Αραβία και να ξέρουμε ότι αν δεν αλλάξουμε τα πράγματα είμαστε συνένοχοι. Υπάρχουν χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν όμως τελικά την Αίγυπτο σε αυτά που κάνει. Ευχαριστούμε. Βόλης. Πρόεδρε, ο πρόεδρος Τραμπ πρόσφατα αποκάλεσε τον αγαπημένο του δικτάτορα τον πρόεδρο Σίση της Αίγυπτας. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αίγυπτο και η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων. Είπα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία ε, κλείνουν τα μάτια απέναντι στα εμπαραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Σίση. Πριν γίνει ο Σίση πρόεδρο, ήταν ο πρόεδρος, μάλλον ήταν αυτός που επέβλεψε μια από τις μεγαλύτερες σφαγέ που έγιναν στη σύγχρονη ιστορία το 2013. Είναι ένας βίος δικτάτορα. Ε, ε, οι Ευρωπαίοι όμως σταμάτησαν να του πουλάνε όπλα. Όχι. Σταμάτησαν να πουλάνε όπλα μήπως του Σαουδάραβε που κάνουν γενοκτονία στην Εμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι δραστικό. Όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει κυρώσεις που είναι ε, σημαντικές για τη Βενεζου... κατά της Βενεζουέλας, της Συρίας, της... του Ιράν, ενώ συνεχίζει να συναλλάσσεται με δολοφόνους. Μα τι συμβαίνει. κυρία Τζούλι Βόρντ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Σεπτέμβριο χιλιάδες διαμαρτυρι... Ε, ε, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Κάιρου, ε, της Αλεξάνδρειας, του Σουέζ, ανταποκρινόμενες σε ισχυρισμούς για διαφθορά του Προέδρου Φατά Χαλσίση. Έκτοτε βλέπουμε να έχουν γίνει φοβερές, φοβερή καταστολή ε, των διαδηλωτών, συλλήψεις 4.500 ανθρώπων, ε, ακόμα και νέων παιδιών, 11 ετών από ό,τι φαίνεται. Ορισμένα παιδιά, αυτά τα παιδιά δεν μπορούν καν να πάνε σχολείο. Οι κρατούμενοι ε, έχουν συλληφθεί με κατηγορίες τρομοκρατίας, παραπληροφόρηση και συμμετοχή σε μια αδειοδοτημένες διαμαρτυρίες. Να θυμίσουμε λοιπόν στην κυβέρνηση της Αιγύπτου ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν τις απόψεις τους και στα κοινωνικά δίκτυα. Ευχαριστούμε αγαπητοί Ε, το λόγο λοιπόν ε, έχει ο Επίτροπος για να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Αίγυπτο. Είναι λοιπόν, ε, είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον ε, γίνεται, υπάρχει πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακριβώ όπω το προβλέπουν οι διεθνεί υποχρεώσει ε, τη χώρα και οι προτεραιότητε που έχουμε καθορίσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο η Αίγυπτος να βελτιώσει την κατάσταση στα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, να βελτιωθεί η ελευθερία έκφραση σε όλα τα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η ελευθερία του συνέρχεσθε, τα δικαιώματα των ακτιβιστών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χαιρετίζει τι τη θέσπιση ενός νέου νόμου για τις ε, ΜΚΟ που αντικαθιστά τον ε, πολλάκις ε, καταδικασμένο νόμο του 2017. Η ελευθερία, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να μπορεί να εργάζεται ελεύθερα και να καταργιστούν όλα τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος των ακτιβιστών. Πολλές συλλήψεις έγιναν μετά τις διαμαρτυρίες του Σεπτεμβρίου του 2020 και δυστυχώς αφορούσαν και πάρα πολλούς που δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Ανησυχεί ιδιαίτερα ότι οι συλλήψεις αφορούσαν πολιτικούς, ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους, ε, Πολλοί εξ αυτών ε, κατηγορήθηκαν ε, με ε, κατηγορίες για τρομοκράτες, παράδειγμα Αλφατάχ, Μοχενούρ, Αλμάση, Αλάμπτελ Φατάχ και ο Μουχάμετ Αλμπάχαλ. Αυτά όλα λοιπόν αντιβαίνουν στο, στις κατάλληλα θετικέ εξελίξεις στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για αναφορές που υπάρχουν για κακομεταχείριση, ε, βασανιστήρια, εξαφανίσεις. Ε, οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως προβλέπεται στις διεθνείς προδιαγραφές. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία για όλες τις μορφές βίας και καταστολής εις βάρος των ακτιβιστών αλλά και πολιτών που προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να διαδηλώσουν ειρηνικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι ε, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκφράζει κανείς ε, αντίθετη άποψη. Η κοινωνία των πολιτών δεν θα πρέπει να εφίστεται μέτρα καταστολής ε, όπως παραδείγματος χάρη είναι απαγόρευση ε, ταξιδιού στο εξωτερικό. Ε, έχουμε διάλογο με την Αίγυπτο στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, κατετέθηκαν έξι τροπολογίες. Η ε, συζήτηση ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα ε, αργότερα, σήμερα το μεσημέρι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η συζήτηση για το προτινόμενο νέο ποινικό δίκαιο στην Ινδονησία και εκλήθη να σας ε, ενημερώσω ότι την μπλε κάρτα μπορείτε να την ανακοινώνετε είτε σηκώνοντα στο χέρι σας είτε ηλεκτρονικά ε, και για τη ε, διαδικασία Catch ε, μπορείτε ήδη τώρα να δηλώσετε ηλεκτρονικά ότι επιθυμείτε να λάβετε λόγο και δεν χρειάζεται να περιμένετε να φτάσει, να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να φτάσει τότε ε, το Catch the Eye. Βεβαίως για να τα κάνετε όλα αυτά πρέπει να έχετε μαζί στην κάρτα σας που να μπορείτε να την τοποθετήσετε στη σχισμή. Περνάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση του θέματος. Οι συντάκτες της έκθεσης ε, έχουν το λόγο και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Άννα Φωτίγκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ινδονησία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντική και για τη δικιά μου τη χώρα, την Πολωνία. Όλες οι ανησυχίες που εκφράζονται στο σχέδιο ψηφίσματος της ομάδας μου, του ECR, τίθενται και στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με την Ινδονησία. Ειλικρινά ζητάω από τους συναδέρφους ευρωβουλευτές να υιοθετήσουν την τροπολογία που υπέβαλα και που έχει να κάνει με έναν Πολωνό, έναν ταξιδιώτη, ο οποίος από λάθο ε, κατηγορείται για προδοσία, για πέντε χρόνια φυλάκιση. Ειλικρινά θέλω να θέσω αυτό το θέμα γιατί πρόκειται για λάθος και το θέτω και εκ μέρους όλων των Πολωνών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρκ είναι επόμενος. Ο κύριος Μπέρκ παρακαλώ. Δεν είναι στην αίθουσα. Δεν είναι στην αίθουσα από ό,τι φαίνεται. ω εκ τούτου περνάμε στον ε, επόμενο ομιλητή Βιλανουέβα Ρουίς. Κυρία Βιλανουέβα Ρουίς. Ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ανησυχητική τάση γιατί γίνονται πιο αυστηροί οι ποινικοί κανόνες. Υπάρχει δίωξη αντιφρονούντων και ποινικοποίηση των διαφόρων ε, ιδεών σε διάφορα σημεία του κόσμου. Σήμερα μιλάμε για την Ινδονησία. Η μεταρρύθμιση αυτή που προβλέπεται στην Ινδονησία ξέρει ποιοι είναι οι εχθροί Μιλάει για ιδέες, ιδέες μαρξιστικές, λενιστικές, μιλάει για μη θρησκευτικέ οργανώσεις, μιλάει για βλαυσιμία, που υπάρχει σαν αδίκημα στη χώρα και ποινικοποιεί επίση και τις γυναίκες οι οποίες προχωρούν σε άμβλωση όπως επίσης και τα άτομα που ανήκουν στην κοινότητα των ΛΟΑΤΙΚ. Είναι μια κατάσταση που βλέπουμε ότι η Ινδονησία δεν έχει ξεκαθαρίσει το, τη σχέση της με το παρελθόν της, με την δικτατορία και έχουμε διώξεις πάνω από δεκατομμύρια ανθρώπων. Είναι από μακριά που μας έρχεται αυτή η δίωξη των αντιφρονούντων. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευράς ε, της Ευρώπης παντού και στην Ευρώπη και στον κόσμο παντού. Μιλάμε για φεμινισμό, μιλάμε για πλουραλισμό, για ελευθερίες, αλλά τα ξεχνάμε όλα αυτά πολύ γρήγορα όταν πρόκειται για το ελεύθερο εμπόριο. Ευχαριστούμε κυρία Τσε. Ευχαριστώ η, η Ινδονησία ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι σημαντικό εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πρόσφατες εκλογές ξεκίνησε ένας νέος πολιτικός κύκλος με κοινοβούλιο και πρόεδρο που θέλουν να ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια. Όμως αυτός ο ποινικό κώδικας είναι πολύ επίμαχος. Χιλιάδες Ινδονήσοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και για να πείσουν για την αναβολή ε, του ποινικού αυτού κώδικα. Και αυτό έγινε ξανά και ξανά. Πιστεύουμε ότι τώρα ήρθε η στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, μετάσχει στη συζήτηση αυτή για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές αρχές. Το ψήφισμα αυτό αναφέρεται στα πιο επίμαχα ζητήματα. Πρόκειται για 20 άρθρα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενισχυτικά, γιατί βάλουν τις γυναίκες, τις ελευθερίες, τις θρησκευτικέ και άλλες, την αντισύλληψη, τις εκτός γάμου σχέσεις κλπ. Έτσι όπως έχει σήμερα το νομοσχέδιο αυτό του ποινικού ε, κώδικα, είναι μια πιστοδρόμηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ινδονησία. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε με τον ιστορικό ρόλο της Ινδονησίας ε, υπέρ του κράτους δικαίου, αλλά να μην δεχτούμε τέτοιες αλλαγές, διακόπτει ο Πρόεδρος. Είχατε ένα λεπτό, είσαστε ήδη στο 1 και 20. Επόμενος ε, ο μιλητής ε, Μαριάν Βιν. I have a problem. Oh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα συνεχίσω στα δανέζικα. Το νέο ποινικό δίκαιο στην Ινδονησία βρίσκεται σε αντίφαση με όλες μας τις αξίες και στρέφεται και κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε, σε ένα νόμο δεν μπορεί να παγιώνεται η διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα που ε, καταπατούνται. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τώρα τροπολογίες ε, που κατατέθηκαν επί του ψηφίσματος. Έχουμε δύο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυλακές της Ινδονησίας. Είναι τραγική η κατάσταση για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά δεν ονοματίζεται κανείς, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα υπευθύνων. Εμείς είμαστε κατά της ε, θανατικής ποινής γενικά όταν όμως ε, πρόκειται για μεμονωμένους ανθρώπους, τότε έχουμε έτσι ένα γενικόλογο ψήφισμα ε, το οποίο εστιάζεται σε κάποια θέματα του ποινικού δικαίου. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ψήφισμα για να απελευθερωθούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους πολλούς Ινδονήσιους που θα αναγκαστούν να συμβιώσουν με το νέο ποινικό δίκαιο. Ε, πρέπει να στηρίξουμε το ψήφισμα, αλλά να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες 4 και 5. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ε, Ο κύριος Σντεχόφσκι. Εν γέννη, Πρόεδρε, μπορούμε να πούμε στο πλαίσιο της ε, Νότιο-Ανατολικής Ασίας ότι η Ινδονησία είναι ένας σταθερός εταίρος. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό και ότι σέβεται κάποιες δημοκρατικές αρχές. Γι' αυτό και μας εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο ότι στη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα που πλέον ε, ε, έχει ολοκληρωθεί, ε, υπήρξαν κάποια σημεία τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν ε, την ανάπτυξη της χώρας αυτής. Και τοποθετεί την Ιδονησία ε, ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες που είναι ακραίες και που παραβιάζει συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και μας χαροποιεί που τους τελευταίους μήνες ο Πρόεδρος διέκοψε την μεταρρύθμιση ε, του ποινικού κώδικα και ξεκίνησε διάλογο με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μορφή της ε, μεταρρύθμισης αυτής, την τελική μορφή. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν και πιστεύω πω έτσι όπω προτάθηκε αυτό ο ποινικό κώδικα δεν θα εγκριθεί. Πιστεύω πω η Ινδονησία θα καταφέρει ακόμα μια φορά να αποδείξει πω είναι σταθερό και δημοκρατικό εταίρο. Ότι είναι ένα εταίρο ο οποίο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια χώρα όπου δεν θα ανανεωθεί η ισχύ της θανατικής ποινή και άλλες καταχρήσεις που αφορούν ε, τις ε, θρησκευτικές μειονότητες. ή άλλου είδους μειονότητες. Πιστεύω πως η διαθεσιμότητα ε, ε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή το ανοιχτό μυαλό, το ανοιχτό πνεύμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα ε, βοηθήσει την Ινδονησία να προχωρήσει θετικά. Μετά λοιπόν τους συντάκτες ε, περνάμε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και στους ε, μεμονωμένους βουλευτές που ζήτησαν τον λόγο. Πρώτα απ' όλους ο κύριος Κέλλη. Καλημέρα σας. Η η Ινδονησία είναι από τις πιο μεγάλες χώρες στον κόσμο, 265 εκατομμύρια, βασικά μουσουλμανική χώρα, αλλά και με μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά τις μειονότητες, τις ρισκίες, τις γλώσσες, τον πολιτισμό. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα η οποία προοδεύει πραγματικά πολύ και είναι μια χώρα όπου μπορούμε να έχουμε στενότερη εταιρική σχέση στο μέλλον. Ως μέλος της Αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ασία και μέλος της Επιτροπής Εμπορίου, ελπίζω πως τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσουμε προς μια ε, μελλοντική ε, συμφωνία συναλλαγών ή εταιρική σχέση με την Ινδονησία. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γιατί ο ποινικό κώδικας για τον οποίο δυσκολευόμαστε εμείς είναι στη διαδικασία κύρωση στην Ινδονησία. Τονίστηκε ότι ως αποτέλεσμα των διαμαρτυριών που αποτρέπονται σε μια λειτουργική δημοκρατία που είναι η Ινδονησία, ο πρόεδρος αποφάσισε να αναβάλει την κύρωση αυτού του ποινικού, νέου ποινικού κώδικα. Άρα λοιπόν τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία, με τα οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι και που δεν ε, ε, ανταποκρίνονται στις διεθνείς σαν διεθνή πρότυπα, δηλαδή δικαιώματα των, μειον, των θρησκευτικών μειονοτήτων, δικαιώματα γυναικών, δικαιώματα ΛΟΑΔΜΑ, πολιτικές ιδεολογίες, αναπαραγωγική υγεία και θανατική ποινή. Και πιστεύω πως θα ήταν θετικό για μας, ειδικά με την νέα επιτροπή, να στείλουμε μια αντιπροσωπεία στην Ινδονησία για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ ίδιος ως εισηγητής για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρσι υποδέχτηκα εδώ εκπροσώπους της Ινδονησίας και συζητήσαμε για το θέμα των Ταμίλ. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να στείλουμε μια αντιπροσωπεία, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να συζητήσουμε τα επίμαχα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσιχοντάρου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που προφέρετε καλά το όνομά μου. Υπάρχουν τρία πράγματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα σχετικά με την Ινδονησία. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος για την βλαυσιμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταδικάσετε κάποιος για τις θρησκευτικέ του ιδέες. Έπειτα, ε, οι διατάξεις κατά των γυναικών και κατά των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων του να μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι καταδικασμένοι επίσης σε θάνατο και αυτό είναι το τρίτο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να καταργηθούν αυτές οι προτάσεις. Έχουν αναβληθεί προς το παρόν, αλλά πρέπει να υπάρξει και μορατόριο όσον αφορά τη θανατική ποινή. Ελπίζω η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λύσει αυτά τα ζητήματα και ελπίζω όλοι οι ευρωβουλευτές να υπερψηφίσουν το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κ. Μοχάμετ. Μιλάω για αυτό το θέμα γιατί έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού ανά τον κόσμο και για το ρόλο που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν από μερικέ εβδομάδε, κύριε την Πρόεδρε, ήμουνα στα σκαλιά του Κοινοβουλίου στι Βρυξέλλε για την Διεθνή ημέρα για την ασφαλή άμβλωση. Έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο και έχουμε αναγνωρίσει ότι οι γυναίκες μπορούν να διέπουν το σώμα τους όπως πιστεύουν αλλά δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Ε, η πρόταση για το νέο ποινικό κώδικα στην Ινδονησία το δείχνει αυτό. Η Human Rights Watch είπε ότι η Ινδονησία και ο ποινικό αυτό κώδικα είναι μια καταστροφή για τι γυναίκε, για όσου πιστεύουν, δεν πιστεύουν, για τι μειονότητε ε, κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει φωνή και πρέπει να την υψώσει. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων δεν πρόκειται να την πετύχουμε ποτέ όσο ο μισός πληθυσμό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του και άλλο μισός όχι. Η ισότητα μεταξύ των δύο φίλων είναι στην καρδιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμεί πρέπει να αγωνιστούμε υπέρ αυτών των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Κούνκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η κυβέρνηση της Ινδονησίας είναι μια πρόταση η οποία ε, παραβιάζει και ε, αγνοεί τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι ελευθερίες των ΛΟΑΔΜ, οι ελευθερίες των θρησκευτικών ομολογιών, οι ελευθερίες αυτές περικόπτονται και Αυτά προς ε, όφελος εκείνων που επιθυμούν να στηρίξουν κάποιους άλλους. Αυτά λοιπόν που διαδραματίζονται στην περιοχή αυτή, όλα αυτά επιδεινώνουν τη σχέση της ε, Ινδονησίας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε στην κυβέρνηση της Ινδονησίας ποια ακριβώς είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι κάθε κυβέρνηση έχει μία θεμελιώδη υποχρέωση που είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα φυσικά επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπέκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ινδονησία για πάρα πολλού ε, ήταν το πρότυπο του φιλελεύθερου Ισλάμ. Δεν ισχύει όμω πια αυτό. Έχουμε παρεμβάσει στη δημοκρατική ελευθερία άποψη ε, και νέε αξιόπινε πράξει, όπω η προσβολή του Προέδρου. Αυτά είναι ε, κάτι καινούριο ε, και όλα αυτά τα ε, καταδικάζουμε και εμείς. Ο ποινικό κώδικας στην Ινδονησία μοιάζει καταρχήν να έχει παγώσει, όμως παρόλα αυτά βάζει πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα. Οι άνθρωποι πλέον στην Ινδονησία δεν έχουν την ελεύθερη μετακίνηση και το θρησκευτικό στοιχείο έχει μπει στην καθαρά προσωπική και ιδιωτική τους χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα υποτίθεται ότι θα πρέπει να προστατεύονται από ένα ε, ισχυρό κράτος. Αυτό όλοι είναι δικαίωμά του. Ε, η κυρία Μέρκελ όμως ε, λέει ότι εντάξει θα έρθουν όλοι αυτοί στην Ευρώπη χωρίς να χρειαστεί να απεμπολίσουν τα δικαιώματά τους. Τι γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέες αξίες, νέες τάσεις και με τον τρόπο αυτό εξελίσσονται παράλληλες ε, κοινωνίες. Οι φιλόσοφοι βέβαια λένε ότι ε, μπορεί να υπάρχει μια πλουραλιστική κοινωνία. Ο Χέγγελ λέει ότι η λύση είναι η δύναμη του πιο ισχυρού. Αυτό όμως είναι ένα καθαρά ε, καθαρό πείραμα. Ο πράσινος, ο Κονμπεντίτ, έχει γράψει ότι όταν συναντιόνται ξένοι πολιτισμοί, ε, απλά αναβάλλεται η σύγκρουση. Η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι σκληρή, είναι φρικαλαία, δεν ε, επιδεικνύει αλληλεγγύη. Αυτή η κοινωνία χαρακτηρίζεται από κοινωνικές ανισότητες και τη χαρακτηρίζει η τάση να δημιουργούνται ε, κοινωνίες ε, και ομάδες ε, που αποκλίνουν η μία από την άλλη. Συνοχή λοιπόν όλων αυτών δεν υπάρχει, χάνονται οι αξίες. Η Ινδονησία δεν είναι κατά κύριο λόγο δικό μας πρόβλημα. Όμως Έχουμε ανθρώπους όπως ο Κονμπεντίτ, ο οποίος επιθυμεί να έχει μια κοινωνία χωρίς κανενός είδους ελεγγύη. Την επιθυμεί διακαώς ο κύριος Κονμπεντίτ αυτή την κοινωνία και για την Ινδονησία και για μας. Αυτά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος ε, Βάιμερς. Ε, Ευχαριστώ. Η πρόταση του ποινικού κώδικα στην Ινδονησία μας παραπέμπει στην απεικιοκρατική εποχή και θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Δυστυχώς δεν σέβεται τους, τα διεθνή πρότυπα και οι τελευταίες τάσεις όσον αφορά τα Ισλαμισμό βρίσκονται μέσα σε αυτήν την νομοθετική πράξη. Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος σαρίας. Υπάρχουν και προβλέπονται μια ολόκληρη σειρά διακρίσεων απέναντι στις γυναίκες, απέναντι στις, εθνοτικές, στις θρησκευτικές μειονότητες, στις σεξουαλικές μειονότητες και φυσικά αυτό ισχύει και για την ε, βλασφημία, για μια ολόκληρη σειρά δε ε, μη Ισλαμικών μειονοτήτων. Ακόμα και μια σειρά χριστιανών διώκονται εκεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ακριβώς να αποσαφηνίσει πού τοποθετείται σε σχέση με την ε, απώλεια ελευθερίας και της αρίας σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κολακούσιτς. Ευχαριστώ αγαπητοί σύντροφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις ε, κυριότερες ε, θρησκευτικές και οικονομικές ε, δυνάμεις στον κόσμο και θεωρούμε ότι μπορούμε να δίνουμε μαθήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο το πώς το κάνουμε είναι λάθος. Εξεργαζόμαστε ψηφίσματα εξαιρετικά αυρά. Και εάν οι χώρε δεν σεβαστούν τα ψηφίσματά μας αυτά, δεν συμβαίνει και τίποτα. Μα αυτό μας βλάπτει. Βλάπτει την αξιοπιστία μας και την ε, επιρροή μας. Πρέπει να εγγυηθούμε την τάξη σε ολόκληρο τον κόσμο και με ξεκάθαρο τρόπο. Πριν, ε, πρώτα λοιπόν ένα ψήφισμα, μετά ειδοποίηση και μετά κυρώσεις που θα πρέπει να είναι συνεπής. Μόνο έτσι θα ξέρει κανείς ότι ε, εάν δεν ε, τηρήσουν τον νόμο θα έχουν συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίζελερ Λίμα. Πρόεδρε, ο νέος ποινικό κώδικας στην ε, Ινδονησία μας οδήγησε σε αυτό το ψήφισμα και μετά από τις διαμαρτυρίες των φοιτητών σε ολόκληρη την Ινδονησία αλλά και στην Δυτική Παπουασία. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν τη στήριξή μα ε, στην αντίθεση στο νέο αυτό ποινικό κώδικα γιατί ποινικοποιεί ό,τι στοιχείο έχει να κάνει με την ταυτότητα του ανθρώπου για την ιδιωτική του ζωή, την ελευθερία σκέψης, την ελευθερία διάθεσης του σώματος του καθενός. Εμείς ε, λοιπόν πρέπει να αντιταθούμε και να υπάρξουν κυρώσεις. Κυρίως γιατί το Σεπτέμβριο θυμόσαστε τι είχαμε ψηφίσει και η Εθνική Επιτροπή που υπάρχει στην Ινδονησία κατά της διαφθοράς φαίνεται να εντάσσεται πια στο κυβερνητικό σώμα, οπότε δεν εξασφαλίζεται η ισότητα όλων απέναντι στον νόμο. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις θετικές σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ινδονησία, εταιρική σχέση, της διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς περιμένουμε πολλά λοιπόν από τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα λάβει η χώρα τον Νοέμβριο φέτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στρουγκαρίου Ραμόνα. Ευχαριστώ πολύ. Στα ρουμανικά θα συνεχίσω, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνία συνεργασίας με την Ινδονησία ήδη από το 2014. Σήμερα έχει αλλάξει η κατάσταση. Έχουμε ένα νέο ποινικό κώδικα που θέλει να αντικαταστήσει τον σημερινό με νέα άρθρα τα οποία παραβιάζουν σαφέστατα τα δικαιώματα των γυναικών, των θρησκευτικών μειονοτήτων, σεξουαλικών μειονοτήτων, την ελευθερία έκφραση και συνεταιρίζεστε. Υπάρχει μια νομοθεσία επίση κατά τη διαφθορά που γίνεται πιο ευάλωτη τώρα. Οπότε λοιπόν ρωτάω, δεν πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε μια νομοθεσία τύπου Μακνίσκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείνουμε τα μάτια δεν μας κάνει συνένοχους στις συνεχείς αυτές καταχρήσεις σε τέτοιες χώρες με τις οποίες όμως έχουμε συμφωνίες συνεργασίας και εμπορικές συμφωνίες. Δεν γινόμαστε συνένοχοι των δικτάτορων αυτών που έχουν τα χρήματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτώ και κάτι ακόμα. Στο ψήφισμα της ομάδας Renew υπήρχε ένα τμήμα για την ελευθερία τύπου ε, για το γεγονό δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να υφίστανται ε, πίεση. Εξαφανίστηκε αυτό όμως το εδάφιο. Γιατί, πού είναι η αλληλεγγύη μας συνάδελφοι. Ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Τρεις έχουν ζητήσει τον λόγο μέχρι τώρα. Και ξεκινάμε με τον κύριο Πόσπισιλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμένα μου αρέσει που όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου πράγματι να μιλάμε για την ε, ποιότητα, την ουσία του ποινικού κώδικα. Γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς έχει κατάσταση σε μια χώρα. Η πρόταση αυτή λοιπόν καταφέρνει να επικρίνει την κατάσταση. Η πρόταση αυτή που υπέβαλε ε, το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας όμως δεν έχει να κάνει με ποινικό κώδικα. Ε, πρόκειται για ρήτρε που ξεκάθαρα παραβιάζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των γυναικών, των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων κλπ. κλπ. Ένας ποινικό κώδικας όταν είναι κώδικας μιας χώρας πρέπει όντως να φροντίζει για το δίκαιο. Ενώ τώρα είναι πολύ ασαφής και μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσει από πλευρά της κυβέρνηση της Ινδονησίας. Γι' αυτό και θέλουμε να απορριφθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζούλι Βόρτ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πάνω από 18 προβληματικά άρθρα μέσα σε αυτό το προτινόμενο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας που μπορούν να περιορίσουν πολλές σημαντικές ελευθερίες. Έχουμε προτινόμενα άρθρα που είναι επιζήμια για τις γυναίκες, για την ομάδα των ΛΟΑΔΜΑ, για τις ε, θρησκευτικές ε, μειονότητες. Υπάρχουν άρθρα κατά της ελευθερίας του λόγου. Όλα αυτά δεν συμβαδίζουν ε, με τις προδιαγραφές της διεθνής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Κανένα κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ρυθμίζει την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων ποιον θα ερωτευτούν, ε, ούτε μπορούν τα κράτη να αστυνομεύουν αποφάσεις ε, των ανθρώπων για το δικό τους το σώμα, παραδείγματος χάνει την ε, αναπαραγωγή των γυναικών. Γνωρίζω ότι η πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση, στην αντισύλληψη, αυτό μπορεί να σώσει ζωές. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τις Ινδονησιακές αρχές να αλλάξουν πορεία και να αφαιρέσουν όλα αυτά τα προβληματικά άρθρα που είναι άρθρα του προηγούμενου αιώνα. Ad hoc ε, ζήτησε το λόγο κυρία Μπάρμπαρα Γκίψον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εξακολουθώ να είμαι και συγκλονισμένη και εννοεί από το γεγονός ότι το 2019 εξακολουθεί να υπάρχει διακριτική μεταχείριση και προσπαθούμε να ελέγξουμε σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι να έχουμε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου ή επίσης να μην αφήνουμε τους ανθρώπους να παντρεύονται. Αυτός ο ποινικό κώδικας βιάζει τα πάντα που εγώ πιστεύω. Πρέπει να σταματήσει. Και χαίρομαι που δείχνουμε αλληλεγγύη για τους ΛΟΑΔΜ, για τις γυναίκες και για όλους τους άλλους που προσβάλλονται, που θίγονται σε αυτή, στην Ινδονησία. Μπότσακ Στάνισλαβ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καταδικάσω αυτό το σχέδιο ποινικού κώδικα στην Ινδονησία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας είναι σταθερός μας εταίρος. Ε, θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις μαζί της. Είναι στρατηγικός εταίρος σε αυτή την περιοχή. Όμως, αν αυτά τα δρακόντια, ο δρακόντιος ποινικό κώδικας και έτσι και πολύ γενικός και αφηρημένος, οφείλουμε να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι οικουμενικά. Δεν πρέπει βέβαια να ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο όπως τα εννοούμε εμείς, αλλά προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ε, παραδείγματο χάρη η δίκαιη δίκη, που είναι οικουμενικά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θεωρώ ότι και η ΝΙΝ και η Μελλοντική Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ αυστηρές και να συζητήσουν με την κυβέρνηση της Ινδονησίας σχετικά με το θέμα αυτό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον Επίτροπο κύριο Μιμίτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, η Ινδονησία μια σταθερή δημοκρατία με ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ, με ζωντανά μέσα μαζική ενημέρωση, έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην θέσπιση ενό νομικού πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση των δημοκρατικών ελευθεριών. Η μακρά διαδικασία εξυγχρονισμού του πεπαλαιωμένου ποινικού κώδικα ε, έφερε θετικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, περιόρισε το φάσμα και τη χρήση της θανατικής ποινής. Ωστόσο, η, η διαδικασία αυτή έχει δημιουργήσει ανησυχίες για διάφορα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει επισύρει κριτικές ε, εγχωρίως αλλά και την προσοχή έχει προκαλέσει τις διεθνούς κοινότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρακολουθήσει στενά στη διάρκεια των ετών την αναθεώρηση του ποινικού ε, κώδικα μέσω τακτικής ε, επαφή με το Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τη κοινωνία των πολιτών και, και διεθνεί εταίρου. Ορισμένε από τι πιο επίμαχε τροπολογίε σχετίζονται μεταξύ άλλων στι διατάξει για την βλασφημία, για την ποινικοποίηση του ε, των εξωγαμιών επαφών και τον περιορισμό των, ανθρωπ... των δικαιωμάτων έκφρασης, των ε, κοινοτήτων ε, ΛΟΑΔΜΟ και των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων. Καλούμε την Ινδονησία τώρα που δεν είναι μόνιμο μέλος αυτή τη στιγμή του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ι.Ε. να τηρήσει τις διεθνεί της υποχρεώσεις και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και να ενεργήσει καταλήλως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλαπλές προσπάθειες ε, για επαφές με τις Ινδονησιακές Αρχές. Για παράδειγμα, το 2018 η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία και τα κράτη-μέλη συναντήθηκαν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και φέτος το καλοκαίρι είχαν επαφές με την αντίστοιχη Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η αφαίρεση του σχεδίου πρόβλεψης ε, ε, που έθετε εκτός νόμου τις ε, σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου. Ε, επίσης, η αναβολή της ψηφοφορίας για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα που παρέπεμψε τη συζήτηση στο νέο κοινοβούλιο το οποίο ανέλαβε φέτος τον Οκτώβριο καθώς και επερχόμενη ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα γίνει ε, το Νοέμβριο στις Βρυξέλλες θα πιέσουμε εκεί την Ινδονησία για τον ποινικό κώδικα και θα θυμίσουμε τις υποχρεώσεις της υπό το Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τα τροπολογίες κατατέθηκαν από διάφορες πολιτικές ομάδες. Η συζήτηση λοιπόν ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα όπως ε, και ε, για όλα τα υπόλοιπα θέματα στις 12 η ώρα. Διακόπτεται προς το παρόν η συνεδρίαση. Presidente. Καλημέρα σας. Ε, αν θέλετε να καθίσετε παρακαλώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Σαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στον Ιαμ Τότι. Ο Ιαμ είναι καθηγητής οικονομίας και είναι και ε, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιγούρων στην Κίνα. Αγωνίστηκε πάρα πολύ για να βελτιώσει την ε, σχέση του κράτους με τους Ιγούρους στην Κίνα και ε, το καθεστώς τον ε, φυλάκισε σε διαβίου φυλακή. Το Κοινοβούλιο λοιπόν επιθυμεί και ζητά να αφαιθεί πάρα αυτά ελεύθερος από τις κινέζικες αρχές. Και μία άλλη ανακοίνωση που έχω να κάνω και αφορά στη σύνθεση του κώδικα συμπεριφοράς των βουλευτών και σε περίπτωση σύγκρουσης οικονομικών συμφερόντων. Α, με βάση τον, ε, τον κώδικα της διοντολογίας αποφασίσαμε να ε, ονομάσουμε Χούπνε, Πισαπία, Μέλχιο, Χάουτολα και Μπουρζουά, να ορίσουμε αυτούς τους συναδέλφους ε, ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την συμπεριφορά των βουλευτών. Και επίσης τους συναδέλφους Άνεμανς και Σόλτς να τους ορίσουμε ως αναπληρωματικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εχθές ε, λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, των Τούρκων βορειοανατολικά της Συρίας ένα μέλος αυτού του κοινοβουλίου συμπεριφέρθηκε με απαράδεκτο τρόπο. Επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, κανένα σεβασμό στους συναδέλφους και κανένα σεβασμό στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι επειδή συμφωνήθηκε και με τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, ότι στο μέλλον δεν θα δεχτώ καμία τέτοια συμπεριφορά που ενδέχεται να ζημιώσει την αξιοπρέπεια και τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. με βάση το άρθρο 166.1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίσαμε να επιβάλλουμε ε, τιμωρία με βάση το άρθρο 13 στον Αντζολο Τσόκα ο οποίος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση είχε μία ε, ταραχώδη συμπεριφορά ε, άφησε τη θέση του και πέταξε κάτι στο κέντρο της αίθουσας. Η κύρωση λοιπόν είναι ότι για 10 μέρες χάνει το δικαίωμα στην ημερήσια αποζημίωση και επίσης ε, προσωρινά αναστέλλεται η δυνατότητά του να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Ε, πέντε μέρες ε, στο Κοινοβούλιο και στις επιτροπές και αντιπροσωπείες. Αυτό από τις 4 Νοεμβρίου βεβαίως χωρίς να αμφισβητηθεί το δικαίωμά του ε, ψήφου στην Ολομέλεια, γιατί έτσι ακριβώς προβλέπεται στον κώδικα συμπεριφοράς των βουλευτών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον βουλευτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει αυτή την απόφαση, να την εφεσιβάλει απευθυνόμενος στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου και κάνοντας χρήση και αναφορά το άρθρο 167. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα που ξεκινάει η κοινοβουλευτική δραστηριότητα, υπήρξαν συμπεριφορές που είναι απόλυτα καταδικαστές, τόσο στον αφορά το, τη γλώσσα όσο και τη συμπεριφορά. Έγραψα κάποιες επιστολές σε βουλευτές και περιμένω την απάντησή τους. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρατεί το πνεύμα της ανεκτικότητας και της ελευθερίας. Όμως η συμπεριφορά και η γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς πρέπει να δείχνει σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μορένο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σα και το κάνω αυτό με μεγάλη συγκίνηση, ένα ιστορικό γεγονό το οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη χώρα μου. Και αυτό είναι η μεταφορά με όλες τις νόμιμες εγγύησεις των γνωστών του δικτάτορα Φράνκο που φεύγουν από ένα δημόσιο μαυσολείο όπου βρίσκονταν μέχρι τώρα και πηγαίνουν σε ένα νεκροταφείο. Παρακαλώ, λίγο σεβασμό. Με την ε, πράξη αυτή η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ τηρεί την υπόσχεσή του και επιστρέφει την ιστορική και δημοκρατική αξιοπρέπεια στην Ισπανία και στους Ισπανούς. Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι είναι μεγάλη δημοκρατία η Ισπανία. Σύγχρονη, ανοιχτή και θέλει να κλείσει μια ιστορία της ιστορίας της, μια τραγική σελίδα της ιστορίας της. Μια στιγμή. Νομίζω ότι σήμερα όλοι οι δημοκράτες πρέπει να ποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα του εμφυλίου πολέμου, του φραγκισμού, ε, στις οικογένειές τους, στις γιαγιάδες μου και στους παππούδες μου και στον πατέρα μου. Κέρδισε η δημοκρατία σήμερα και βρισκόμαστε στον οίκο της δημοκρατίας εδώ. Grazie. E adesso Non è un dibattito. E adesso procediamo alle votazioni. Προχωράμε τώρα. Ε, προχωράμε στο θέμα των ΛΟΑΔΜ στην Ουγγάντα. Παράγραφος 4 με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. La votazione è chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα, πάντα με ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε παρακαλώ για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στο ψήφισμα από πέντε πολιτικές ομάδες για την Αίγυπτο, παράγραφος 14, υπέρ παρακαλώ, να ψώσετε το χέρι, κατά, αποχές, επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτό. Παράγραφος 16. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Παρακαλώ να ψώσετε το χέρι. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος, μάλλον, ε, τροπολογία 2, παράγραφος 16, ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το ε, αιτιολογία 1, το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές ε, παλήθευση παρακαλώ έκλειση ψηφοφορία δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται μετά το εκτιμώντας έχουμε την τροπολογία 1 ε, ψηφίζουμε παρακαλώ με ονομαστική κλίση Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, δεκτό το ψήφισμα. Πάμε τώρα στην ε, πρόταση για τον ποινικό κώδικα στην Ινδονησία. Ε, μετά την παράγραφο 3, τροπολογία 3, ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε παρακαλώ, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8 σε 4 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ε, δεκτό. Τρίτο τμήμα, ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτό. Votazione è aperta. Εγκρίνεται λοιπόν. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1, παράγραφο 9, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ανομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες του σύνολου, του συνόλου μάλλον. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Ομαρζή. Έχουμε μόνο μία ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ κύριο Μαρζέ. Εκτός. Εκτός μικροφώνου. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο αυτό. Ε, χρησιμοποιήστε το διπλανό αν θέλετε. Α, εκώ, εκώ, Α, τώρα λειτουργεί. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 4, τέταρτο εδάφιο του κανονισμού, ζητάω ως πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής το θέμα αυτό να επιστραφεί στην Επιτροπή Ρέγγι εν ώψη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ψηφίζουμε την πρόταση του κύριου Μαρζέ. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνονται. Άρα λοιπόν παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Τώρα, ε, ένσταση για την... Ε, ε, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι για τη μερική χορήγηση άδεια για μια χρήση του διοξιδίου του χρωμίου. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Conseguenze del fallimento del gruppo Thomas. Τώρα, ε, επιπτώσεις της χειροκοπίας του ομίλου Thomas Cook. Τροπολογία 8. Νομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Για διαδικαστικό στο 18, στον κατάλογο Τόμας Κούκος, στο δεύτερο εδάφιο, το ΕΛΚ έχει κάνει λάθος και πρέπει να βάλουμε συν εκεί στον κατάλογο ψηφοφορία δηλαδή του ΕΛΚΑ. Παράγραφο 10. Per alzata di mano. Παράγραφο 10. Διανατάσσω ότι ισχυρό Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπο... Ε, παράγραφος 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18 σε 6 τμήματα. Ένα, πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Έγκρινεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Έκτο τμήμα. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας J, αρχικό κείμενο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, πληροφορίες για το φόρο εισοδήματο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βορειοανατολική Συρία συνέπειες. Τροπολογία 3, παράγραφος 2, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Παράγραφος 3. Άρχεται. Απορρίπτεται. Παραγραφός 4. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. 12. Τροπολογία 12. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 10. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8, με ονομαστική κλίση. Άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική κλίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην επόμενη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι δύο υπέρ, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα σχετικά με τη Μεσόγειο, πρόταση ψηφίσματος του ECR. Ε, ψηφίζουμε για το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται το ψήφισμα. Πάμε τώρα ε, στην πρόταση ψηφίσματος της ομάδας e D. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα του ΕΛΚ στο σύνολό του. Υπέρ, παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα, πρόταση ψηφίσματος ε, της Επιτροπής ε, για τις Πολιτικές Ελευθερίες, ε, παράγραφος 1, η τροπολογία 41. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42D. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρθών 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεκτή. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. δεκτή η τροπολογία. Καταπίπτει λοιπόν το αρχικό κείμενο, τροπολογία 43D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 44 και 59 ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται τροπολογία 60D ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία Απορρίπτεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 45 δι με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε έκλειση ψηφοφορία απορρίπτεται η τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 46 υπέρ ψηφίζουμε ψηφίζουμε Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 21D και 47D και 61D ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 29 τροπολογία. 29 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 48. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 49. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 22. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 62. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 77. Υπέρ παρακαλώ. Έκλειση ψηφ... Αντίθετα, ε, αποχή, ε, επαλήθευση, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 2 καταπίπτει. Τροπολογία 63D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Όχι, μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Τι έγινε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 23 με ανάταση χειρός υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 78 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 64 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Η 50D. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 65 πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 51D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 66 πρώτο Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 52 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 53D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 67. Υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή. Η 79. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Η 80 πρώτο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 54. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 68. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Η τροπολογία 69 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 70. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. 71. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. 72. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 56D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά. Η 56 τώρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 15, 26D και 57D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, δυστυχώς πρέπει να κάνουμε παλήθευση. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα καταπίπτει, το δεύτερο καταπίπτει. Πάμε στην 58D τροπολογία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται. Η 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή καταπίπτει το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 30. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 4. Υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 28. Υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 5. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας C, ε, τροπολογία 6, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 8, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 31. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 31. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 74. Υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή. Η 32. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 9. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 10D και 33D ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Η τροπολογία 34D, το εκτιμώντας L, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας M, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 35D απορρίπτεται. Εκτιμώντας ο, ο. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε παρακαλώ. έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 36 ψηφίζουμε παρακαλώ. έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 12. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 30, 13D και 37D ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Η 38D ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η 15D υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 39 ψηφίζουμε παρακαλώ. Η 39. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 16D και 40D. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τώρα ψηφίζουμε για το ψήφισμα. Στο σύνολό του ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του απορρίπτεται. Passiamo Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, έναρξη προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Πρόεδρος Λόπες Αγγιγιάρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνο για να πω ότι είναι μια μέρα που πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το θάνατο 39 ανθρώπων οι οποίοι ήταν θύματα ε, σωματεμπορίας. Τέτοιοι θάνατοι λαμβάνουν ε, χώρα στους δρόμους, στη Σαχάρα αλλά και στη θάλασσα. Συνεπώς, για λίγες ψήφους δεν μπορέσαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Όχι μόνο σε αυτούς που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αλλά για να δείξουμε τη στήριξή μας σε ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να σώζει αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Γιγιάρα. Θα περάσουμε στην έναρξη πρωταξιακών διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Πρόταση ψηφίσματος από 6 πολιτικές ομάδες, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15, πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Ζετόφσκι. Όχι. Ναι, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχω μια σύντομη προφορική ε, τροπολογία. Τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την άρνηση της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Και για τη διεύρυνση. Και αυτό είναι ε, αρνητικός αντίκτυπος στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν αυτή η πρόταση. Υπάρχουν αντίθετοι. Οι αντίθετοι ποιοι είναι. sono ci sono anche loro? Sì, sono più di 40. Bene. Sì, sì, sì. Quindi, sì. Quindi passiamo avanti. Όχι, λοιπόν, περνάμε. Ε, προχωράμε. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πάνω σε αυτή την προφορική. Λοιπόν, παράγραφος 2, παρα, ε, τροπολογία 16 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το πρωτότυπο κείμενο. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Πρωτότυπο κείμενο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 15 ε, άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται 8 δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας α άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται εκτιμώντας β άρχεται πέρας εγκρίνεται εκτιμώντας ε τροπολογία 10 ε, συγγνώμη Ι λοιπόν είναι τροπολογία 10 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Περ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύνολο της, ε, του ψηφίσματος τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Grazie. Buon rientro e grazie della collaborazione. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Διακόπτω για λίγα λεπτά. Παρακαλώ, σιγά σιγά σας ζητάω όσοι θέλετε να βγείτε από την αίθουσα να βγείτε ησύχως και οι υπόλοιποι που παραμένουν να μπορέσουν να μιλήσουν και να παρουσιάσουν την επεξήγηση ψήφου τους. Okay. Akkor Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτο σημείο είναι οι επιπτώσεις της πτώχευσης της Thomas Cook. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Χάουαρτ, εκ μέρου των ε, Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κατάρρευση της Thomas Cook έχει σοβαρές επιπτώσεις στους υπαλλήλους αλλά και στις επιχειρήσεις και στον τουρισμό παντού στην Ευρώπη. Πρόκειται για 21.000 πελάτες οι οποίοι περιμένουν να αποζημιωθούν για τα ταξίδια αυτά που έχασαν και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το Catwick που είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο για τσάρτερ στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, βλέπει να χάνονται ε, Πολλέ θέσει απασχόληση που εξαρτώνται από τη Thomas Cook. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να ζητήσει να αναλυθεί ενδελεχώ η πτώχευση αυτή και να δούμε τι θα μπορούσε να αποφύγει τέτοιε καταστάσει στο μέλλον. Το ψήφισμα επίση τονίζει και τι δυνατότητε που δίνονται από το Ταμείο για την Αντιμετώπιση τη παγκοσμιοποίηση για να προστατευτούν αυτοί που χάνουν τι δουλειέ του και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διευκόλυνση για να βοηθήσουμε πραγματικά αυτού που ψάχνουν δουλειά τώρα και γράφω στο Γενικό Γραμματέα και του ζητάω όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πάλμερ. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν θα κατέβω απόψε από το τρένο στο Λέστερ, θα δω το άγαλμα του Τόμας Κουκ, που έχει υψωθεί για να τιμήσει την μνήμη του, την επιχείρηση και κάποια από τα πρώτα ταξίδια που οργάνωσε το 1885. Πρώτο οργανωμένο ταξίδι στην Ευρώπη που περιελάμβανε τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Και βεβαίως οι επιβάτες ε, σε αυτά τα ταξίδια ε, δεν θα είχαν την, ε, την προστασία του συνδέσμου ΑΤΟΛ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να φροντίσουμε όσοι επηρεάζονται από τέτοιες καταρρεύσεις ε, σήμερα να προστατεύονται πλήρως ε, στο μέλλον και να αντληθούν τα κατάλληλα διδάγματα από την κατάρρευση της ε, Thomas Cook που επηρέασε 600.000 πελάτες και πολλούς χιλιάδες εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπελαμή. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Μα είμαστε σοβαροί βουλευτές ψηφίσαμε ένα ψήφισμα σήμερα για τον Τόμας Κούκ και για την Τουρκία. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. εκπλήσωμε για τα ψηφίσματα εδώ πέρα και τις ψηφοφορίες μας. Έχουμε λύσει δηλαδή όλα τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τα προβλήματα των άλλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται και οι ευρωβουλευτές με το να δίνει παραδείγμα στον υπόλοιπο κόσμο. Και νομίζουμε ότι είναι σήμερα το χθες. Θέλουμε να στηρίξουμε κάποιες αξίες. Πώς όμως ε, ε, παρεμβαίνουμε στο εσωτερικά χωρών και ε, δημιουργούμε εντάσεις, ιδίως αν πρόκειται για κράτη-μέλη της Ένωσης. Τόσο ότι φοβόμαστε τη δημοκρατία σε κάποιες χώρες όπως η Πολωνία και δεν τους αφήνουμε να λύσουν εκεί με το δημόσιο διάλογο τα εσωτερικά τους ζητήματα. Το δικαίωμά μας είναι να πούμε και όχι. Ε, θέλουμε να υπηρετούμε το καλό, την ε, ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Ε, όχι να ελέγχουμε τι κάνουν οι άλλοι. Τελικά φλιαρούμε και καθιστάμεθα ανίσχυροι. Μέχρι τελικά να νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα εικονικό δικαστήριο και όχι σε ένα κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ έχει τώρα το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε ε, παρόντες για να βοηθήσουμε μετά από την ε, τρομακτική ε, πτώχευση του ομίλητο Μασκούκ. Καταναλωτές, ε, πελάτες, επιχειρήσεις ε, έχουν πληγεί πολύ από αυτή την υπόθεση. Αλλά τα κράτη-μέλη ουσιαστικά έχουν την ευθύνη και δεν μου αρέσει που η αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου προσπαθεί να εμπλέξει την Κομισιόν. Περισσότερο από όσο θα έπρεπε στο θέμα αυτό. Με διάφορες προτάσεις. Για μείωση παραδείγματο χάρη των πόνους. Ε, μα αυτό θα το αποφασίσουν οι μέτοχοι. Είναι θέμα ιδιωτικού δικαίου. Δεν νομίζω ότι η δημόσια ε, ε, εξουσία έχει να δραματίσει κάποιο ρόλο εδώ. Δεν έχει να κάνει δηλαδή εδώ με θέσει περί και Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τώρα. που είναι η κατάσταση που σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματο αφορισμένε επιχειρήσει και υποκαταστήματα, δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις αιτιολογήσεις ψήφου για την έκθεση αυτή με πρώτη την κυρία Σκοτ Κέιτο. Όταν οι πράσινοι εδώ πέρα ζήτησαν να αναφέρονται δημοσίω τα κέρδη των τραπεζών του 2015, φώναζαν οι τράπεζε ότι θα χρεοκοπήσουν, αλλά μια χαρά τα πάνε. Το να έχουμε δημόσιε πληροφορίε για το πώ μεταφέρουν τα κέρδη του είναι ο μόνο τρόπο να διασφαλίσουμε ότι θα πληρώνουν φόρου. Γι' αυτό αντιστέκονται αλλά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν πρέπει να τους βοηθούν. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για, την, για το εταιρικό δίκαιο θα συνεδριάσει αύριο για το θέμα αυτό. Φαίνεται πως η γερμανική θέση με αλλάζει και το καλωσορίζω. Αν και λυπούμε για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παίξει ρόλο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν στο Συμβούλιο για να υπάρχει διαφάνεια στις επιχειρήσεις. Εάν έχει κάποιο νόημα η ευρωπαϊκή συνεργασία, ακριβώς σε αυτόν τον τομέα πρέπει να φανεί. Γιατί και οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με μεγάλες που φοροδιαφεύγουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Πόσπισιλ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως εισηγητής για το συγκεκριμένο θέμα με χαρά επιβεβαιώνω την άποψη ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα η διαφάνεια στο θέμα το φορολογικό, ιδιαίτερα στα πλαίσια της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Η αλήθεια είναι ότι στο Συμβούλιο όμως υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Η Φιλανδική Προεδρία είπε ότι θα προσπαθήσει να μετακινήσει κάπως το Συμβούλιο. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Η θέση του Κοινοβουλίου ε, νομίζω είναι σαφής και σταθερή. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της τεχνικής βάσης, αλλά αυτό είναι τεχνικό. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρειο-ανατολική Συρία. Η επίθεση της, Συρίας, της, της Τουρκίας συγγνώμη, στη Βόρεια Συρία παραβιάζει τις αρχές του, δι, του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αγνοούμε τα συμφέροντα των Κούρδων που ήταν οι σύμμαχοί μας στην καταπολέμηση του Ντάες. Τώρα το Ντάες έχει πιθανότητες να επανέλθει. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μας σύνορα. Χτυπήσαμε κατά τη διάρκεια της ε, Ουκρανικής κρίσης στη Συρία. Και τώρα η Τουρκία εισβάλλει στη Συρία και δεν υπάρχει καμία αντίδραση θα πρέπει να σταματήσουμε να δίδουμε επιστώσεις στην Τουρκία. Ό,τι έχει σχέση με την προενταξιακή βοήθεια και με το πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση πρέπει να διακοπούν. Θα πρέπει επίσης σε πολυμερές επίπεδο να υπάρξει μια διεθνή συνάντηση για το Συριακό με συμμετοχή της κυβέρνησης της Δαμασκού. Ευχαριστώ πολύ. Jones, ευχαριστώ πολύ. Μάλλον ε, πρόσφατα ξεκίνησε η Τουρκία μία ε, θανατηφόρα επιχείρηση. Υπάρχουν ε, αποτροπιαστικές πράξεις βάρος άμαχου πληθυσμού. Ε, και απελευθέρωση πολλών τσιχατιστών μαχητών. Να καταδικάζονται όλα αυτά από τα κρατημένα. μπορούσε όμω να υπάρχουν ε, να είχαν επιβληθεί οικονομικέ κυρώσει ε, μετά από την επίθεση και ενώ η Άγκυρα εκβιάζει με μεταναστευτικό την Ευρώπη, θα μπορούσαν οι Βρυξέλλε να είχαν τερματίσει οριστικά τη διαδικασία ένταξη με την Τουρκία που ούτε από πλευρά αξιών, ούτε πολιτισμού, ούτε γεωγραφία ανήκει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε όμω. Δίνουμε δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Η τροπολογία μας ε, απορρίφθηκε από 542 βουλευτές ε, ε, που είναι ουσιαστικά η συνένοχη της Τουρκίας και μεταξύ αυτών και το Ανμάρς του Μακρόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ψήφισμα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην ε, Βορειοανατολική Συρία ε, είναι σωστό διότι καταδικάζει την τουρκική εισβολή, ζητά να την ε, πάυση, τον τερματισμό της και την απόσυρση όλων των Τούρκων από τη Ρωσάβα. Υπενθυμίζει ότι η δαυκή κυριότητα, η κυριαρχία τη Συρία πρέπει να γίνουν σεβαστέ, όπω και το δικαίωμα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών συνιστοσών τη χώρα. Γι' αυτό και στηρίζω αυτό το ψήφισμα. Θα πρέπει όμω να πηγαίνει λίγο πιο μακρά και να καταδικάζει απερίφραστα το θάνατο ε, του Σεριν Καράφ, καθώ επίση να ζητά ε, την ανάπτυξη ειρηνευτική ε, δύναμη ε, και ανώκρανων για την προστασία των Κούρδων ε, και για να να δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση εντό του Συριακού κράτου. Ε, πρέπει να μην ξεχνάμε του Κούρδους που είναι σύμμαχοί μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Πόσπισιλ έχει τώρα τον λόγο. Από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ στήριξα αυτό το ψήφισμα. Πιστεύω ότι η Τουρκία παρανόμως ε, επιτίθεται στους Κούρδους ε, της Συρίας. Δείχνει ξεκάθαρα πως η Τουρκία δεν προσεγγίζει την Ευρώπη, μάλλον απομακρύνεται. Από αυτήν τα έχουμε πει πολλές φορές. Και βεβαίως ε, δεν έχει πλέον νόημα να μιλάμε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συζητηθεί του εάν θα παραμείνει και μέλος ε, του ΝΑΤΟ καθώς η πολιτική της αντιστρατεύεται το ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. είναι ο κύριος Χόρβουντ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την εντονότερη δυνατή καταδίκη της εισβολής ε, και το να βλέπουμε Ερντογάν και Πούτιν να μοιράζουν τα ημάτια της ε, Συρίας ε, ενώ συγκατανεύει ο Τραμπ είναι τραγική εικόνα. Η ευθύνη νομίζω ανήκει σε μεγάλο μέρος στον πρόεδρο Τραμπ που πρόδωσε τους Κούρδους συμμάχους. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση υψώνει το αναστημά της σε έναν επικίνδυνο κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύουν συνεχώς και οι σύμμαχοί μα, όπως είπα, αποδεικνύονται αναξιόπιστοι. Είναι σαφές λοιπόν πως 28 ε, χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να μιλούν με μια δυνατή φωνή σε ζητήματα εξωτερικής πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ζάχαρα από το e Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία θα πρέπει να καταδικαστεί. Και είναι θετικό αυτό το οποίο προτείνει το, η, το, το ψήφισμά μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι από τη μία μαύρα και από την άλλη λευκά. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι εμείς υποστηρίζουμε κάποιες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να οδηγήσουν στην διάλυση μιας άλλης χώρας. Αυτό θα ήταν απαράδεκτη παρέμβαση στα εσωτερικά της Τουρκίας. Θα πρέπει επίσης να παραδεχτούμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένας παγκόσμιος εταίρος παίκτης πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από το να ψηφίζει τέτοιου είδους ψηφίσματα και να κατηγορεί τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι δεν στέκονται στο ύψος των υποχρεώσεών τους. Διάβασα τη δήλωση Τραμπ χτες και νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν με αυτό. Είπε ότι δεν είναι δουλειά των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων να καταστούν οι χωροφύλακες της παγκόσμιας σκηνής είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και Ρώσοι είναι να αρχίσουν να κάνουν αυτά τα οποία τόσο καιρό λένε. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο θάλασσα. Επεξηγήσεις ψήφου. Η κυρία Σόιντροβα ξεκινάει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Εγώ δεν υποστήριξα το ψήφισμα αυτό, όπως επίσης και κάποιες από τις τροπολογίες. Βέβαια, η τροπολογία τελικά πέρασε από την αρμόδια επιτροπή με δύο ψήφους διαφορά δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε οικονομικούς μετανάστες. Ξέρω ότι ο αριθμός των ε, ΜΚΟ έχουν καλές προθέσεις. Προσπαθούν να διασώσουν τον κόσμο. Αλλά πρώτα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Και θα πρέπει επίσης σε περιπτώσεις κρίσεων να μπορούν να φιλοξενηθούν με καλές συνθήκες σε στρατόπεδα προσφύγων και αν υπάρχουν κάποιοι πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς προστασίας πρέπει να το έχουν αυτό με νόμιμο τρόπο. Νομίζω ότι το να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς ανακατανομής είναι λάθος τρόπος. Έχει απορριφθεί από πολλές χώρες μέλη και δυστυχώς καλύπτει τους οικονομικούς μετανάστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλμερ από το Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το ψήφισμα αυτό καταψηφίστηκε με δύο ψήφους διαφορά. Είναι μια μαύρη μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, ναι. Θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι διακινητές, ναι. Αλλά το θέμα αυτό είναι και απλό, θεωρώ εγώ, γιατί κατ' ουσίαν το θέμα είναι το αν υποστηρίζουμε την ιδέα του να σώζουμε παιδιά που πνίγονται στη θάλασσα, γονείς, παιδιά που κάνουν επικίνδυνα ταξίδια για να αποφύγουν διώξεις και πολέμους. Θέλω λοιπόν οι ψηφοφόροι μου να ξέρουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, πως εγώ υπερψήφισα την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο και το να οδηγηθούν οι διακινητές δικαιοσύνη και να μην ποινικοποιούνται όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Και ψήφισα για μέτρα τα οποία τελικά καταλήγουν σε μια αίσθηση ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο κύριος Μπροντίνσκι για το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι η ψήφος μου συνεισέφερε με τρόπο απτό και το ψήφισμα αυτό καταψηφίστηκε. Δεν ξέρω πως ακούγονται πολλά πράγματα για από αυτό το θέμα, συναισθηματικά. Ένα είδος δηλαδή ηθικού εκβιασμού και ε, μπορεί να νομίζει η κοινή γνώμη ότι συνέβη κάτι το κακό. Όχι, καταφέραμε να καταψηφίσουμε ένα ψήφισμα που ενθάρρυνε εκατομμύρια ανθρώπους να πάνε στην ακτή Λιβύη στην Ισία Μαρόκου και από εκεί να προσπαθήσουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό ε, σήμαινε ότι θα προωθήσαμε Τη ΜΚΟ και τα οργανωμένο έγκλημα. Ήμουν υπουργό εσωτερικών ε, στην Πολωνία, έχω δει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Οι ομάδες αυτές ε, βγάζουν περισσότερα λεφτά από αυτή την υπόθεση από ότι από το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Σας ευχαριστώ. Ντιλ ε, από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ καταψήφισα και χαίρομαι ιδιαίτερως που απερίφθη. Ας τα πούμε τα πράγματα ανοιχτά. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αποτελεσματικά και να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη διακίνηση, τους διακινητές που μεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία, περνώντας ψηφίσματα που όχι μόνο δεν σταματούν ε, τους διακινητές, αντίθετα τους ε, εξαιρεθίζουν περισσότερο για να συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια και περισσότερα. Είχαμε την περίπτωση της ε, καπετάνισσας ε, Καρόλα Ρακέτε που υποτίθεται ότι έσωζε ανθρώπους στη θάλασσα αλλά παρεύει το δίκαιο της θάλασσας και παραβίασε διάφορους κανόνες και ε, θα τιμωρηθεί κιόλας από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να ανακοπούν οι ροές της μετανάστευσης, αλλά όχι να οθούμε τελικά με τα ψηφίσματά μα στους διακινητές να συνεχίζουν το έργο τους. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ενάρξη ανταξιακών διαπραγματεύσεων με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Κυρία Σόιντροβα είναι η πρώτη από το Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εξηγήσω γιατί εγώ στήριξα το ψήφισμα αυτό του Ευρωκοινοβουλίου που επικρίνει τη στάση Ολλανδών, Δανών και Γάλλων. Κυβερνήσεις τους μπλόκαραν την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας και κατ' εμέ αυτό αποτελεί μέγα στρατηγικό σφάλμα. Σίγουρα θα ήταν μακροχρόνιες και πολύπλοκες οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν για να έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική οι χώρες αυτές, οι πολίτες των χωρών αυτών, ότι χρειάζονται την ευρωπαϊκή προοπτική. Πρόσφατα η Βόρεια Μακεδονία συμφώνησε για το όνομά της με την Ελλάδα. Ήταν ε, σημαντική, μια σημαντική συμφωνία και ε, να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χάσει ε, την ε, επιρροή που μπορεί να ασκήσει. Και δεν είναι καλό το ότι θα πάει στην Σερβία. Ευχαριστώ κυρία Κιόβεβα να σας εξηγήσω γιατί υπερψήφισα εγώ αυτό το ψήφισμα για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Γιατί ε, λόγω ενός κράτους μέλους ε, διακυβεύεται το μέλλον ολόκληρης τη περιοχής. Δεν δέχομαι τη γαλλική θέση, όχι μόνο επειδή η χώρα μου, η Σλοβενία και η Βόρεια Μακεδονία ανήκανε κάποτε στη Ιουγκοσλαβία. Η μάνα μου είναι από εκεί. Εγώ λοιπόν έχω απογοητευτεί προσωπικά ως άνθρωπος που γνωρίζει τι είναι να σου υπόσχονται κάτι επί σειρά ετών, να κάνεις ό,τι σου ζήτησαν και στο τέλος τίποτα. Λοιπόν, το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα είναι ένα μήνυμα ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία πάνε προς σωστή κατεύθυνση και οι δύο χώρες γνωρίζουν ότι έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Βεβαίω Ε, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ε, ακόμα απέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλάμε για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρουτζίνσκι από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Βόρειας Μακεδονίας άκουσε αυτά τα οποία συζητήσαμε χτες και δυστυχώς ακούστηκαν πράγματα τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι οι εκπρόσωποι των μεγάλων κρατών βλέπουν με απέραντη περιφρόνηση τους εκπροσώπους των μικρών χωρών μια σλαβικής χώρας όπως η Βόρεια Μακεδονία. Αυτό μου θυμίζει αυτό το οποίο έλεγαν παλαιότεροι ιστορικοί σε σχέση με το Βοναπάρτη. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έκανε ο πρόεδρος Μακρόν. Δεν είναι ένα απλό λάθος, είναι ένα βαρύ λάθος. Αν ήξερε τι σκέπτεται ο λαός της Βόρειας Μακεδονίας, δεν θα είχε λειτουργήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Τσόρτσιλ είχε πει για τα Βαλκάνια πράγματα πολύ σημαντικά τα οποία αγνοούμε. Η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία έχουν καταστήσει πλέον τα Βαλκάνια μια πυρητιδαποθήκη με εξτρεμιστές από τη Ρωσία και από τη Σαουδική Αραβία στην Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Τσάχραντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και υπεψήφισα την πρόταση αυτή γιατί προέρχομαι από αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Μία περιοχή η οποία ε, εδώ και 15 χρόνια μόνο αναγνωρίστηκε ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό οι χώρες μας δεν έχουν κανένα ηθικό δικαίωμα ε, να ε, καταδικάζουν ορισμένες χώρες και να μην δέχονται τις, ε, την ένταξή τους στην Ένωση. Πέραν τούτου θα πρέπει να κατανοήσουμε γιατί επίσης ορισμένοι από τους γείτονές μας είναι σχετικά διστακτικοί σε σχέση με την, με την περαιτέρω διεύρυνση. Κάποιες παλιές χώρες διστάζουν και πιστεύουν ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει να κάνει με την Ανατολική Ευρώπη. Αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία και στην Πολωνία περιπλέκουν τα πράγματα. Πρέπει να δείξουμε κατανόηση και αν το κάνουμε τότε θα αλλάξουμε και την άποψή μας. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, μετά από τις τελευταίες παρεμβάσεις διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι την, ε, τρίτη, την, τις 3 το μεσημέρι. Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα χθεσινά πρακτικά και το κείμενο που υιοθετήθηκαν είναι διαθέσιμα και ε, εγκρίνονται. Το σημείο που έχουμε υποσυζήτηση είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή ε, για τον ε, τοποθέτηση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ Φάρκας, του κ. Φάρκας, ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME. Να σας πω ότι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τη στάνταρ εγγραφή και το νέο σύστημα που επιτρέπει στα μέλη να εγγραφούν ηλεκτρονικά για μπλε κάρτες. Σας καλώ λοιπόν να φέρνετε πάντοτε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας. Αν θέλετε λοιπόν να εγγραφείτε για το Catch the Eye, σας καλώ να το κάνετε τώρα, χωρίς να περιμένετε για το τέλος της συζήτησης. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση και θα δώσω το λόγο στο συντάκτη, τον κύριο Τάνκ. Έχετε το λόγο. Yes. Thank you, Mrs. President. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ επίσης για την διαδικασία Catch the Eye που μας ενημερώσατε. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο Άνταμ Φάρκας, που είναι εκτελεστικός διευθυντής της CDA, θα γίνει και διευθύνων σύμβουλος της ΑΦΜΕ. Είναι αξιοσημείωτο. Είναι εντυπωσιακό και αποστομωτικό ότι ο εκτελεστικός διευθυντής αυτού του τομέα ε, στην ουσία μετατρέπεται στο βασικό λομπίστα για τον τομέα αυτό η EDA θεσπίζει τους τραπεζικούς κανονισμούς και τους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν οργανισμός για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και είναι στόχος το όλων των λόμπι, ειδικά της ΑΦΜΕ με την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που εστιάζει στα εφαρμοστικά μέτρα τα οποία συντάσσει η EDA και έχει διαρκή ε, επαφή με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξή μου όταν έμαθα ότι ο εκτελεστικό διευθύντη τη εποπτική Αρχής θα γίνει διευθύνων Σύμβουλο τη της ε, ε, ε, ΑΦΜΕ που είναι ένα τραπεζικό λόμπι, έχει ειδική πρόσβαση στο υψηλότερο ιστάμενο προσωπικό. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ε, επηρεάσει υπερβολικά βασικές, βασικά νομοθετήματα. Επιπλέον, αυτό που είναι χειρότερο είναι ότι μπορεί να δώσει την εντύπωση στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη λάθος ιδέα ότι δηλαδή αν είσαι φιλικός προς έναν οργανισμό θα αμυφθείς ε, ε, με μια υψηλά αμοιβόμενη θέση οι κανόνες της Ένωση πρέπει και θέλουν να το εμποδίσουν αυτό. Το άρθρο 16 του εστερικού κανονισμού ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι ε, υπάλληλοι ε, ε, απαγορεύεται να ασκούν πίεση σε προσωπικό του πρώην οργανισμού τους για μια περίοδο ενός έτους. Το να διατηρεί δηλαδή τέτοιο επαφή στην ουσία σημαίνει ότι ακυρώνει την περιγραφή του, της θέσης απασχόλησης. Πώς θα γίνει δηλαδή ο ίδιος να μιλά με τον εκτελεστικό, το μέλλοντα εκτελεστικό διευθυντή του ίδιου του οργανισμού του Πιστεύουμε πως έτσι βλάπτονται τα θεμητά συμφέροντα αυτού του θεσμού. Η χρηστή εποπτεία του τραπεζικού τομέα δεν είναι ο στόχος αυτής της αρχής. Αυτό υποσκάπτεται από την κίνηση του Φάρκας. Αν αυτή η υπόθεση περιστρεφόμενης πόρτας δεν οδηγεί σε επαρκή, ε, ε, σε, μάλλον, δεν οδηγήσει σε επαγόρευση αν επιτραπεί κάτι τέτοιο, οποιοδήποτε Ευρωπαίος υπάλληλο θα επιτρέπεται να μπει σε τέτοιες θέσεις και καθ' θα καταστεί το άρθρο 16 άνευ Εχθές ξεκινήσαμε μια ε, αναφορά με ε, πολλούς συναδέλφους κατά αυτής της υπόθεσης. Πολλοί αισθάνονται μεγάλη απόγνωση και οργή. Εξ ονόματος λοιπόν των πολιτών της Ευρώπης σας ρωτώ, θεωρείτε ότι η κίνηση φάρκας είναι σύμμορφη με τα υψηλά ηθικά πρότυπα των ευρωπαϊκών οργανισμών. Συμφωνείτε ο κύριος Φάρκας να παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Θα θα ασκήσετε πίεση στην EBA να αλλάξει τη θέση της και να παρεμποδίσει αυτή την επαγγελματική κίνηση του κύριου Φάρκας. και τι ακριβώς θα κάνετε ώστε να θέσετε σε, να μετατρέψετε σε πράξη τα πρότυπά σα και τα πρότυπά μας, ώστε να μην υποβαθμιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμού μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Επιτροπό Μίμτσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών από τον ίδιο τον κανονισμό της είναι υποχρεωμένη να τηρεί ένα πλαίσιο διοντολογίας όσον αφορά τις διάφορες θέσεις. Και το πλαίσιο αυτό αφορά και περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τοποθέτηση του προσωπικού σε άλλες θέσεις μετά από την σταδιοδρομία του στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Υπάρχει και σώμα το οποίο είναι υπεύθυνο για τις ε, αποφάσεις όσον αφορά αυτούς ακριβώς τους περιορισμούς. Οπότε, όσον αφορά τον κύριο Φάρκας, τέτοιες ε, προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να τοποθετηθεί στη νέα του θέση. Ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ψηφίζουν στο σώμα εποπτείας. Όμως, ο κύριος Φάρκας είναι και μπορεί να συνεισφέρει σε σε αυτό το Συμβούλιο. Συνεπώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε όσο γίνεται πιο αυστηρά να προσεγγίσουμε το θέμα της αποχώρησης του κύριου Φάρκας, λαμβάνοντας υπόψη μας τον κανονισμό του προσωπικού. Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσον αφορά τους περιορισμούς για τον κύριο Φάρκας, όταν αποχωρήσει, έγιναν ε, γνωστές. Υπάρχουν περιορισμοί όσο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Πρόκειται και για μέτρα που καλύπτουν ένα χρόνο κοινοποίηση για να γίνει γνωστό που θα τοποθετηθεί μετά. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν πάυση κάθε δραστηριότητας που έχει να κάνει με την προετοιμασία του ρυθμιστικού, της ρυθμιστικής ή της εποπτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Τραπεζών, την εξωτερική της ε, εκπροσώπηση και πληροφορίες εκτός αυτής. Οι περιορισμοί συμπεριλαμβάνουν και τρεις μήνες περίοδο κατά την οποία δεν ε, ε, φέρει σε πέρα στον ρόλο του ρυθμιστή ή εντελοδόχο και δεν μπορεί να βρίσκεται στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εκτός να το ζητήσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αυτό το τρίμηνο. Τώρα όσον αφορά την αποχώρηση, για την περίοδο μετά την αποχώρηση. Το Συμβούλιο Εποπτών αποφάσισε ότι ο κύριος Φάρκας δεν μπορεί να ασχοληθεί με λόμπινγκ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ούτε μπορεί να έχει επαφές με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για 24 μήνες. Δεν μπορεί να συνεισφέρει στο έργο οργανώσεων που ασχολούνται με το χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Ευρώπη ούτε με κάτι που έχει σχέση με τα καθήκοντά του τα τελευταία τρία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και αυτό για 18 μήνες. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί για να, υπάρχει, να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από την, την περίοδο κοινοποίηση μέχρι την αποχώρηση αλλά και μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και είναι ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να θέσει σε εφαρμογή όλου αυτού του περιορισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Φερνάνδης έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια για να έχει κανείς εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σύμφωνα με τις έρευνες, διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα και αυτή η μειωμένη εμπιστοσύνη ε, χρησιμοποιείται από τους λεκιστές για να υπονομεύσουν όχι μόνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά και τις ίδιες τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Συνεπώς, η είδηση αυτή εξόδου του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και η μετάβασή του σε ένα από τα πιο σημαντικά λόμπι της Ευρώπης συνεισφέρουν ακριβώς σε αυτήν την ιδέα που έχει ο κόσμος για το ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σκέφτονται δηλαδή οι πολίτες ότι οι υπάλληλοι, το προσωπικό, οι πολιτικοί δεν εξυπηρετούμε τους λόγους για τους οποίους βρισκόμαστε εδώ. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να καθίσουμε και να σκεφτούμε τι σύστημα ελέγχου διαθέτουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ένα σύστημα βάσει του οποίου εκείνοι οι οποίοι εργάζονται και συνεργάζονται με αυτούς που θα φύγουν από ένα όργανο για να πάνε αλλού είναι πιο κατάλληλοι για να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Μα δεν έχει νόημα αυτό. Και εδώ δεν θα καθίσω να συζητήσω την εφαρμογή της ρύθμισης. Αυτό που συζητάω και λέω είναι ότι η ρύθμιση δεν έχει κανένα νόημα και ότι πρέπει να έχουμε ένα ανεξάρτητο όργανο, ένα ευρωπαϊκό ανεξάρτητο θεσμό, ο οποίος θα αξιολογεί κατά περίπτωση τέτοιες ε, περιπτώσεις. Γιατί αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τα θεσμικά όργανα και πηγαίνουν σε λόμπις, δεν μπορεί να έχουν αλλιώς ανεξάρτητο κριτήριο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση για την αναθεώρηση των κανόνων. Ευχαριστούμε τώρα εκ μέρου των πράσινων για τρία λεπτά ο κύριος Καρέμ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και ο συνάδελφος, η σύγκρουση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να διαρκέσει άλλο, γιατί αυτό υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στη Γαλλία είναι εθνικό σπορ. Ο Μακρό δούλευε στην τράπεζα πριν να γίνει υπουργό και μετά πρόεδρος, ε, αλλά μας λένε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχουν να κάνουν με τα δώρα που γίνονται στους πιο ε, επιτυχημένους ούτε ότι υπάρχει σύγκρουση φερόντων με το πυρηνικό, με το πυρηνικό όμιλο ε, Αρεβά σήμερα. Επίσης ε, έχουμε τον ε, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος προσελήφθη από την τράπεζα Goldman Sachs. Σήμερα ακόμα μια εξοργιστική υπόθεση εκεί όπου ο κύριος Φάρκας ήταν διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που προσπαθεί με νύχη και με δόντια αποφύγει επίσημη άλλη κρίση ε, μετατρέπεται σε διευθύνων σύμβουλο της ΑΕΦΜΕ, η οποία αυτό που θέλει να κάνει να μην περάσει καμιά άλλη νομοθεσία σχετικά με τις τράπεζες, να εμποδίσει την υιοθεσία άλλης τράπεζας. Είναι ένα από τους κεντρικά, κεντρικούς όμιλους λόμπινγκ ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα αυτός. Επίσης, ε, είπατε ότι 24 μήνες θα απαγορεύεται να ασκεί λόμπι στο προσωπικό του προηγούμενου του θεσμού ή ακόμα πιο απίθανα απαγόρευση για 18 μήνες να συμβουλεύει να εργάζεται για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την προηγούμενη του θέση. Μα ποιος το πιστεύει όλα αυτά και κυρίως ποιος μπορεί αυτό να τα επαληθεύσει και πώς δεν θα κάνει λόμπι όταν έχει στοιχεία ε, ε, πολύτιμα και ε, απόρριτα που θα χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή η κατάσταση είναι σκανδαλώδης και δεν θα πρέπει να επιτραπεί. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς οι κανόνες σε θέματα τέτοια μέσου θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει χώρος για υποψία σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ε, θα πρέπει να ορίζουμε πολύ πιο μακρές περιόδους μετάβασης ανάμεσα σε δύο θέσεις απασχόλησης όπου πιθανά δυνητικά να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην ορίζουμε περίπτωση και ένα οργανισμό. Ε, τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την ηθική και τη διοντολογία. Θα είναι υπεύθυνη για να υποπτεύει του κοινού αυτού κανόνε, αλλά αναμένοντα αυτό θα μπορούσαμε ήδη να δράσουμε σε επίπεδο του δικού μα θεσμού για να προστατεύσουμε την ακαιρεότητά του ενάντια σε αυτέ τι σκανδαλώδει πρακτικέ. Γι' αυτό προτείνω, όπω το Κοινοβούλιο το έχει ήδη κάνει για του λομπίστε τη Μονσάντο, να αρνηθούμε την πρόσβαση του κυρίου Φάρκα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα για να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε ε, πια ε, καταλάβει ότι πρέπει να πάψει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στα μεγάλα αφεντικά και τις ομάδες συμφερόντων. Δύο λεφτά τώρα, ο κύριος Ρουίθ Ντεβέσα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, ακόμα και αν δεν είναι και καλύτερη ώρα, ούτε η καλύτερη μέρα, γιατί πολλοί από τους συναδέλφους μας ήδη έχουν φύγει μετά από τις ψηφοφορίες, αλλά πάντως ε, πάλι καλά και επίσης ε, να χαιρετήσω την ε, παρουσία πολιτών στα θεωρία. Τους χαιρετίζω γιατί είναι ζήτηση μεγάλης σημασίας όπως τόνισαν και οι συνάδελφοι της ομάδας, ο κύριος Τάγκ και Φερνάντες, τους οποίους συγχαίρω που υπέβαλαν αυτή την προφορική ερώτηση και ο συνάδελφος και φίλος Καρέμα από τους Πρασίνους. Γιατί πραγματικά βρισκόμαστε ενώπιον τουλάχιστον μιας ε, υποψία σε σύγκρουση συμφερόντων και ξέρουμε ότι θα πρέπει όχι μόνο να είμαστε αλλά και να φαινόμαστε αλλά και να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, ε, σε αυτή την περίπτωση έχουν ε, χρησιμοποιηθεί πολύ ευνοϊκοί όροι για τον κύριο Φάρκα, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει κανεί, όπω είπε ο συνάδελφο, ότι ε, λέμε ότι απαγορεύεται να δώσει καμιά συμβουλή για θέματα τα οποία σχετίζονται με την προηγούμενη του θέση. Δεν λύνει το πρόβλημα, διότι όπω είπαν και οι συνάδελφοι προήμουν από μένα, δικαίω είναι στην πράξη αδύνατο να επαληθευθεί αυτό, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι και να δίνει πληροφορίε για την προηγούμενη του θέση χωρί να υπάρχει καμιά απολύτως δυνατότητα να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και εγώ χαίρομαι που η Κομισιόν με τη δική της ψήφο σε αυτό το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ζήτησε την εφαρμογή, την αυστηρή των κανόνων, αλλά είναι προφανές ότι αυτό δεν αρκεί. Οι κανόνες θα πρέπει να καταστούν ε, πιο αυστηροί, αλλά και η εφαρμογή αυτών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί μια υποχρεωτική μετάβαση τουλάχιστον 12 μηνών στον κύριο Φάρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα για τρία λεπτά ε, και πάλι ο κύριος ε, Τάνκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή ε, για την απάντηση που μας έδωσε. Αυτά μας που μας ε, είπατε δεν μας πείσανε γιατί αναφέρατε τις ε, προϋποθέσεις που συνοδεύουν την μεταπίδηση του κυρίου Φράγκας. Και εγώ σας λέω ειλικρινά αυτά δεν μας ικανοποιούν. Αναφέρατε τη δυνατότητα να μην δεν τότε τότε στο Φάρκας να έχει το συμβόλαιο αυτό με την ΕΑΤΑ αλλά κατ' ουσίαν ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο επαγγελματικό. Δηλαδή η ΑΤ αναφέρει ότι ο κύριος Φάρκας ε, δεν μπορεί να συμβάλλει σε θέματα που έχουν άμεσα σχέση με τη δουλειά που έκανε τα τελευταία τρία χρόνια. Και αυτό το βρίσκω πραγματικά αστείο. Ε, δεν μπορώ να σκεπτώ ούτε ένα θέμα που να καλύπτει ο κύριος ε, Φάκας που να μην έχει σχέση με τη δουλειά του. Και γι' αυτό λοιπόν ρωτώ και πάλι. Ο κύριος Φάρακας θα βρίσκεται ε, στον πύργο της ΕΑΤ ε, δεν θα δουλεύει σε κάτι σημαντικό και τελικά ποιος θα ελέγχει ε, κατά πόσον ο κύριος Φάρκας συμμορφώνεται με τους περιορισμούς της ΕΑΤ όπως είπε και ο κύριος Φερνάντας. Ποιος θα διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αυτοί οι περιορισμοί. Και ακόμα χειρότερο, ο κύριος Φάρκας θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην ΕΑΤ μέχρι την αναχώρησή του. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνη και παρόλα αυτά η ΕΑΤ ζητά από τον φορολογούμενο να πληρώσει για την πολυτελή μεταπίδησή του. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και τέθηκε αυτό από την απάντηση σας κύριε Επίτροπε. Δεν άκουσα να θέλετε λιγάκι να ε, εξαφανίσετε, να καταργήσετε αυτή τη μεταπίδηση των στελεχών του Μπαρόζο και άλλων ε, γιατί φαίνεται ότι δεν λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα και επιτέλους πότε θα εφαρμόσετε τους κανόνες, ε, πότε επιτέλους ε, ε, θα εξαφανίσετε, θα καταργήσετε την αχίλιο πτέρνα που έχει σχέση με την ακεραιότητα του θεσμού που εκπροσωπείτε. Μία, ένα μόνο αίτημα για το Catch the Eye στον κύριο Μπράιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όταν ένας, ένα ανώτατος τέλεχος μια σημαντική τράπεζα ε, ε, βρίσκεται στη θέση του και διαπραγματεύεται με την άλλη πλευρά, ε, νομίζω ότι τότε έχουμε μια εικόνα ότι ο άνθρωπος αυτός εξαγοράζεται φεύγει και εξαγοράζεται. Έτσι και αλλιώ ο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν νιώθει μεγάλη εμπιστοσύνη και εδώ προκαλείται η εντύπωση ότι υπάρχει σύνδεση με στα στελέχη, τα ανώτατα στελέχη των τραπεζών. Ε, υπάρχει δικτύωση και δεν γνωρίζουμε τελικά ε, πότε ξεκίνησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Μήπως ξεκίνησαν όταν ήταν ήδη ενεργό μέλος και μήπως ε, επηρέασε τη δουλειά που έκανε. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πράγματι είναι σωστό να υπάρχει μία περίοδος αδράνειας, να μην ε, προκύπτει καν η υποψία σύγκρουση συμφερόντων. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά αν πιστεύετε ότι ο κανονισμός προσωπικού δεν αρκεί για να επιβληθεί μια τέτοια περίοδος αδράνειας, μήπως σκοπεύετε να προτείνετε μεταρρύθμιση αυτού του κανονισμού προσωπικού. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, και πάλι στον ε, Επίτροπο, στον κύριο Μιμίτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, σημαντική συζήτηση που είχαμε για την προφορική ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι οι ηθικές προδιαγραφές τίθεται σε εφαρμογή καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και σε όλους τους οργανισμούς εφόσον υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή αυτή, και εδώ μιλάω και εκ μέρους και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα λάβει υπόψη την σημερινή συζήτηση που έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κοιτάξουμε και πάλι τις ρυθμίσεις διοντολογίας. Είναι πράγματι ευθύνη του Συμβουλίου του Εποπτικού της Ευρωπαϊκής, Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών τουλάχιστον με το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο να αποφασίζει για τις προϋποθέσεις βάσει των δικών της κανονισμών. Και είναι επίσης αρμοδιότητα πάλι του Συμβουλίου του Υποπτικού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να ελέγχει και να φροντίζει για την εφαρμογή αυτών των ε, κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Τα πρακτικά αυτή τη συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ έγκριση στην επόμενη αρχή συνόδου και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια αυτή θα παραδοθούν στον προορισμό τους. Εδώ διακόπτεται η σύνοδος και λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ.